Αγαπητοί συνάδελφοι, γεια σας. Να ξεκινήσουμε τη συνάντησή μας την απογευματινή. Παρακαλώ όχι συζητησούλες μεταξύ σας. Α, καλό αυτό. Στο σημείο 1 που είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης ε, της 5 Απριλίου μας το είπε η γραμματεία αλλάξαμε τη σειρά των σημείων, του σημείου 5. Είναι η δημογραφική αλλαγή και οι συνεπίε για τη μελλοντική πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κυρία Σάγια που συντάκτη ο άλλαξε η σειρά με το 9. Είναι η πέμπτη έκθεση της Επιτροπής για τη Συνοχή και τη Στρατηγική σχετικά με την πολιτική της συνοχής μετά το 2013. Δεν ξέρω αν κάποιο θα ήθελε μια κάποια παρατήρηση να κάνει. Όχι, εγκρίνεται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στις ανακοινώσεις Προέδρου. Έξι ανακοινώσεις. Μεταδίδεται μέσω ίντερνετ, όπω συνήθως γίνεται. Δεύτερη ανακοίνωση. Μετά ψηφοφορία τη 16 Μαρτίου και αυτό στην Επιτροπή απασχόληση ο πρώτο τρίμε διάλογο για την έκθεση του κ. Κάστλερ για το ευρωπαϊκό έτος αγώνα για το active aging για το, για το ενεργό γύρας λοιπόν από τις 7 ε, παρατέταρτο θα σας ενημερώσουμε ε, για τις ε, διαπραγματεύσεις αυτές. Σύμφωνα με τον κανονισμό μας ε, πάμε τώρα τη τρίτη ανακοίνωση, η προφορική ερώτηση και πρόταση ψηφίσματος για τη Σύμβαση της Διεθνής Γραφείου Να σας πω ότι στους συντονιστές τι κάναμε. Επεξεργαστήκαμε ένα συμβαστικό κείμενο και για την προφορική ερώτηση και για την πρόταση ψηφίσματος. Επίσης, Για τα δύο αυτά κείμενα έχουμε πέντε τροπολογίες που έχουν κατευθεί και 61 για την πρόταση ψηφίσματος και έτσι εάν εγκριθούν ε, τα πάντα θα ξεπεράσουμε έτσι αυτές τις δυσκολίες που μας, ε, θα μας εμπόδιζαν να το υποβάλλουμε αυτό στην Ολομέλεια. Εντάξει, έχουμε το συμβαστικό κείμενο των συντονιστών θα είχαμε και μόνο. Τέταρτη ανακοίνωση. Στους φακέλους σας τι έχετε. Την έκθεση της γραμματείας, η μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας είχε μεταβεί στη Νέα Υόρκη, στην Ηνωμένα Έθνη το Φεβρουάριο που μας πέρασε. Πάμε στην επόμενη ανακοίνωση. Επίσης τους φακέλους σας θα βρείτε κάτι ακόμα. Η γραμματεία μας, η αγαπητή, τα σύνταξε όλα αυτά. Μια ανταλλαγή απόψεων Ένα σημείο ακριβώ για την ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπου των ε, κοινωνικών εταίρων και των μη κοινωνικών οργανώσεων για το ρόλο και τις, ε, τα αποτελέσματα, πώς επηρεάζει τα πράγματα το κοινωνικό ταμείο και από το, έχουμε στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά το σημείο με αυτό. Επίσης δύο νέοι συνάδελφοι, απόντες όμως τώρα, γι' αυτό θα τους ανακοινώσω επίσημα όταν θα έλθουν. Πάμε στο σημείο 3 της σημερινής σας διάταξης, συνέγκριση των πρακτικών της συνεδρίας της 15-16 Μαρτίου του 2011, χωρίς παρατήρηση, άρα λοιπόν εγκρίνονται τα πρακτικά αυτά. Πάμε παρακάτω στο σημείο 4 δηλαδή, οι συμβαστικές τροπολογίες στην έκθεση Ρισάρτ Φάλμπρ για την εξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής, την προώθηση των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και την κοινωνική ευθύνη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο, αλλά ε, κυρία Μωρέ, κάτι θα ήθελα να πει, διαδικαστικά μάλιστα. Ακούστε κυρία Πρόεδρε. Στις ανακοινώσεις σας κανονικά ήταν ε, συμπεριλαμβάνονταν. Ε, δεν με είδατε να σηκώνω το χέρι μου. Παρακαλώ προσέξτε κάτι. Στην περιφερειακή πολιτική, στην επιτροπή αυτή, είχαμε τρεις παραγράφους ε, που συνέταξε η Επιτροπή αυτή η Περιφερειακή και που έχουν να κάνουν με την ευθύνη της δικής μας, τη δική σας Επιτροπής. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είμαι αντίθετη στην πρακτική αυτή και θα ήθελα να αντιδράσετε εξ ονόματός μας όλων μάλιστα. Με συγχωρείτε που σας διάκοψα. Όχι, όχι, όχι, εντάξει στο, δεν το λησμόνισα, το πρόσεξα και ξεκίνησα ήδη τις απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσουμε να το αλλάξουμε αυτό και η κυρία Μπάστος που είναι και η συγγετριά μας για την πέμπτη έκθεση για την συνοχή κοινωνική και τη στρατηγική σχετικά με αυτή. Έχουμε μια συμφωνία όπως πρέπει ακριβώς με την Επιτροπή αυτή, με αυτό το περιεχόμενο. Κύριε Μάισνερ. θα ήθελα να μιλήσω μετά από τον κύριο Φάλμπερ, γιατί εγώ είμαι σκιωδής εισηγήτρια. Μου δώσατε κάπως νωρίς το λόγο, λοιπόν. Κύριε Κάζα, μήπως κάτι θα θέλετε να θίξετε. Ναι κύριε Πρόεδρε, δεν κατάλαβα πολύ καλά αυτό που είπατε σε σχέση με την ε, ε, με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και τις τροπολογίες που συνδέονται με αυτές. Νομίζω ότι το ψηφίσουμε αύριο αυτό το θέμα. Ναι. Μήπως μπορείτε να το εξηγήσετε καλύτερα. Ναι, θα το εξηγήσω με βραδύτερους ρυθμούς, λέει η κυρία Περές. Αύριο θα ψηφιστούν όλες τροπολογίες. Τι γίνεται ίσως γίνει διπλάσιο το κείμενο του ψηφίσματος. Τι προτείνει η Επιτροπή. Πρόταση ψηφίσματος μετά από την προφορική ερώτηση στην Ολομέλεια και προβλέπει ο κανισμός μας, μην με ρωτάτε τώρα το γιατί και με ποιο τρόπο, αλλά τι προβλέπει λοιπόν ο κανισμός μας, ότι μπορούμε να έχουμε μόνο 1500 στοιχεία ανασελίδα και μέχρι 4 σελίδες λοιπόν να ενωθετήσουμε όλες τις τροπολογίες οι οποίες έχουν κατευθεί και οι οποίες είναι 61 μην τα ξεχνάμε, τότε θα διπλασιάσουμε την έκταση του κειμένου, τουλάχιστον του επιτρεπόμενου. Στη συνάντηση των συντονιστών επεξεργαστήκαμε ένα συμβαστικό ακριβώς κείμενο. Το έχετε επίσης στους φακέλους σας για την απόψινή μας συνεδρίαση. Παρακαλώ ρίξτε μια ματιά προσεκτικά ο κ. Σαμπαουρή συντονιστή συμμετείχε στη συνάντηση αυτή και πάνω σε αυτό το κείμενο συμφωνήσαμε. Τι σημαίνει. Ορισμένοι που κατέθεσαν τροπολογίες τις απέσυραν όπως εγώ παραδείγματο χάρη, ενώ άλλοι, εάν θεωρούν ότι το σημείο του είναι τόσο σημαντικό και δεν καλύπτεται όπως πρέπει με τη συμβαστική αυτή λύση που επεξεργάστηκαν οι συντονιστές, τότε θα μπορούσαν να βασιστούν ακριβώς την ψηφορία στην Ολομέλεια για να την επαναπροτείνουν. Εντάξει, απάντησε το ερώτημά σας, ναι. Δεν υπάρχει νομίζω κάτι άλλο. Η εισηγητής, λοιπόν έχει το λόγο και τον ευχαριστούμε για την υπομονή με την οποία μας άκουσε μέχρι τώρα, μέχρι να ξεκινήσει. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Και αυτό γιατί στις προηγούμενες συνεδριάσεις μας είχα την ευκαιρία να εκφράσω τη θέση μου σε σχέση με την έκθεση αυτή, τη θέση μου επίσης σε σχέση με τις τροπολογίες και σε ό,τι αφορά και τις συμβιβαστικές λύσεις. Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει μαζί με τη Βερόνικα να συμφωνήσουμε για τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Μόνο μία τροπολογία της κυρίας Μάισνερ εγώ απέριψα και επιμένω στην απόρριψη αυτή. Αν υπερψηφίσετε τη θέση μου, δεν πειράζει και πάλι ολυμπιακό. Euh, για να δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να εκφράσω την θέση μου. Είχαμε συζητήσει με τον κύριο Φάλμπρο για αυτές τις προτάσεις συμβιβασμού, εγώ εξ ονόμα της ομάδος Άλντε και ε, εδώ αναφερόμαστε στη συμβαστική τροπολογία G στα λατινικά. Αυτή μπορούμε να τη δεχτούμε. Εκεί που έχουμε πρόβλημα είναι η συμβαστική τροπολογία F, σίγμα ταφ, στα ελληνικά. Γιατί εμείς θέλαμε να υπάρξει μια ισότιμη μεταχείριση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους εργαζόμενους και τις ανάγκες να τονίσουμε την οικονομική επιτυχία και την ανταγωνιστικότητα. Νομίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια εξισορρόψη έναντι των δύο αυτών μεριμνών και η τροπολογία, η συμβιβαστική τροπολογία F ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποδυναμωθεί προς όφελος της ανταγωνιστικότητας και των οικονομικών ε, κερδών. Αυτό για μένα αφαιρεί το εξισορροπημένο χαρακτήρα και επομένως έχουμε προβλήματα με τη συμβαστική αυτή τροπολογία F. Ναι, μεν έχει καλύψει την ε, αρχική μας τροπολογία, αλλά όχι με τη μορφή που θα θέλαμε εμείς και έχουμε δυσκολία. Προσπαθήσαμε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε με τον κύριο Φάλμπρα, δεν τα βρήκαμε και επομένως γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε δυσκολία στο σημείο αυτό. Κατά τα άλλα, με ενοχλεί λιγάκι, κυρία Πρόεδρε, που είπε ο εισηγητής ότι δεν μπορούσε να δεχτεί όλες τις τροπολογίες. Φυσικά θα ψηφίσουμε για όλες τις τροπολογίες. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να καταθέσει μία τροπολογία για τα θέματα αυτά. Εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι όταν έχει κάποιος ένα κείμενο, έχει ο κάθε βουλευτής το δικαίωμα να παρουσιάσει τις τροπολογίες που θέλει. Δεν θέλω λοιπόν να μακρηγορήσω, απλώς θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιο όριο σε μήκος στο αρχικό κείμενο όταν έχει τροποποιηθεί. Νομίζω ότι το αρχικό κείμενο περιορίζεται στους 1500 χαρακτήρες και όχι το τροποποιημένο. Δίκαιο, απόλυτα έχετε. αλλά ίσως μια κάποια μικροσύγχυση επικρατεί γιατί αυτός ο περισμός δεν είχε να κάνει με αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης που είχα αναφέρει αλλά σε μία από τις ανακοινώσεις για την πρόταση ψηφίσματος που ακριβώς θα ζητήσουμε στην Ολομέλεια εμείς σαν Επιτροπή αλλά για τις τροπολογίες της για την έκθεση του κ. Φάλου θα κάνουμε το σύνηθες. Δηλαδή πρώτα απ' όλα θα ψηφίσουμε τις συμβαστικές λύσεις. Από τη στιγμή που θα υιοθετηθούν θα καταπέσουν οι τροπολογίες τις οποίες εκείνες συμβαστικές καλύπτουν από τη στιγμή δε που δεν θα υιοθετηθούν θα ψηφίσουμε σήμερα με τη σειρά του προβλήθηκε ο μας τις 10 τροπολογίες αντίστοιχες. Κύριε Φωτόγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα Ο κύριος Πάρα πολύ, πάρα πολύ σύντομα θέλω να αντιδράσω, Το να ψάχνουμε μια ισορροπία με κάθε τίμημα είναι ο δρόμος που στρώνει την οδό, είναι, στρώνει το δρόμο για την κόλαση. Δεν ξέρω αν πρόκειται για βιβλική έκφραση, αλλά που θα πρέπει να καθοδηγεί και την συζήτησή μας. Ε, κύριε Φοντάγια, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που ακριβώς ε, άκουσε και δέχτηκε πολλές συμβαστικές τροπολογίες. Καταλαβαίνω βέβαια και ορισμένε αφελίες που τρέφει ε, σε αυτό ε, που διατηρεί και κάποιο τόνο κριτικό, εντάξει, και που νομίζω ότι είναι για όλους μας θετικό. Επίσης, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι εάν εγκρίνουμε αυτή την ε, έκθεση που όπως ελπίζω καταλαβαίνουμε ότι η προστασία των δικαιωμάτων εργαζομένων δεν είναι εκείνη που όπως θα έπρεπε να είναι σε αρκετές χώρες όπως και σε αρκετά κρατημέλη, σε κρατημέλη αλλά και μερικές φορές ακριβώς τις ε, συμβάσεις ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας δεν, δεν σέβονται. Να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή της οικονομικής κρίσης όπως υποφέρουμε επίσης ε, δεν θα πρέπει δεν μπορούμε να λέμε όχι στο ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο που έδωσε ήδη καλά θετικά αποτελέσματα. Δεν ξέρω μήπως θα ήθελε να κάνει κάτι για την τροπολογία ο εισηγητής, ε, για την τροπολογία αυτή, για το κοινωνικό ε, ευρωπαϊκό πρότυπο και φιλελεύθεροι να μπορέσουν να ψηφίσουν. Εντάξει, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά επαναλαμβάνω, οπωσδήποτε θα πρέπει να, ψηφιστεί, να, πρέπει να διατηρηθεί αυτό το πρότυπο το δικό μας το κοινωνικό το ευρωπαϊκό. Επίσης για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τους υπόλοιπους συναδέλφους γιατί νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα θετική αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φοντάνια. Τι σημαίνει αυτό. Εντάξει, ως έχει αυτή την εύτολο το λατινικό μπορείτε να την ε, υποστηρίξετε αυτή την ε, συμβαστική Κυρία Στανούκα, ποιος είναι μετά, ποιος είναι... Ας αρχίσουμε την κυρία Στανούκα. Yes, thank you. I'm a shadow Ευχαριστώ. Είμαι Σκιώδης εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Φάλμπερ για την ελαστικότητα, για την ευελιξία που επέδειξε. Η συνάντηση που είχαμε στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ιδιαίτερα καρποφόρα. Ε, αποφασίσαμε για διάφορες τροπολογίες και οι τροπολογίες της ομάδας μας συμπεριλήφθηκαν. Ιδιαίτερα στη συμβαστική Α και στην F, σίγμα και στην G, Z. Οπότε, καταρχήν, στηρίζουμε την γραμμή του εισηγητή. Κάποιες μικρές διαφορές υπάρχουν όσον αφορά την οργάνωση, ε, διεθνή οργάνωση εργασίας και στη συμβιβαστική σίγμα ΤΑΦ που λέει ότι η Επιτροπή ζητάει συνεργασία και δίνει κάποια παραδείγματα εκεί. Ελπίζω οι συνάδελφοι να τα υποστηρίξουν. Οπότε συγχαρητήρια στον κύριο Φάλμπρο. Ευχαριστώ. Τσίμαρ και μετά Μόραν. Ευχαριστώ. Και εγώ από τη δικιά μου την πλευρά και για τη δικιά μου την ομάδα πρέπει να πω ότι στηρίζουμε γενικά μιλώντας, την ε, γραμμή που ακολουθεί ο εισηγητής. Νομίζω ότι με τους συμβιβασμούς, τις συμβαστικές ε, τροπολογίες δηλαδή, μπορούμε τελικά να συμφωνήσουμε. Στις διαπραγματεύσεις που έγιναν για τις συμβαστικές τροπολογίες, ε, προσπαθήσαμε να πάνε αυτές όσο γίνεται πιο μακριά. Και αυτό ώστε να συμφωνούν με τον κανονισμό και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην υπάρξει αποδυνάμωση των κειμένων. Η θέση του Ευρωπαϊκού του Κοινοβουλίου έτσι βελτιώνεται πιστεύω. Θα έλεγα μάλιστα ότι η συμβαστική τροπολογία F σιγματάφ είναι μια τροπολογία που μπορούμε να στηρίξουμε. Δεν μπορούμε όμως να δεχτούμε επιπλέον αποδυνάμωση της τροπολογίας αυτής. Συμφωνούμε πάντως με το σύνολο του κειμένου. Ευχαριστώ. Κύριε Μωράν, για να... παίρνω το λόγο για να σας πω το εξής. Χτες με τον Αλεσάνδρο Σέρκας στην μόνιμη ομάδα εργασίας με τα συνδικάτα ε, συζητήσαμε μαζί τους και δουλέψαμε νομίζω πάρα πολύ καλά πάνω στην ε, έκθεση αυτή. Από πλευράς του ΕΛΚ είμαστε υπέρ όλων των συμβαστικών τροπολογιών, γιατί εκεί συμπεριλαμβάνονται οι δικές μας ε, τροπολογίες και χαιρετίζω το έργο των σκιωδών εισηγητών, διότι χάρη σε αυτό καταφέραμε να φτάσουμε σε τέτοια θετική σύγκληση πάνω στην έκθεση αυτή που είναι πολύ σημαντική για την πρόοδο της κοινωνικής Ευρώπης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Άλλος? Α, ήξερα ότι κάποιον ξέχναγα. Ο κύριο Τόμα Μάν έχει το λόγο. Συγγνώμη, ήξερα ότι κάποιον ξέχναγα. Να. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ σίγουρα δεν νιώθω ότι είμαι αντικείμενο διάκριση. Είμαι στον κατάλογο των ομιλητών. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ήθελα να πω ευχαριστώ στον Ρίτσαρτ για αυτά τα οποία έχει κάνει. Αν έχει καταφέρει κανείς από 155 διαφορετικές τροπολογίες να βρει μια συμβιβαστική ε, θέση, αυτό δεν οδηγεί στην κόλαση όπως είπε, μπορεί να μην οδηγεί και στον ε, παράδεισο βέβαια, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θετικό βήμα και έχει βοηθήσει όλους μας. Και εγώ είδα και από την πλευρά των σκιωδών εισηγητών πόσο θετικό είναι να μπορεί κανείς να καταλήξει σε κοινές θέσεις. Λοιπόν, η κόλαση είναι για μένα ο χώρος εκεί που δεν υπάρχει καμία συμβιβαστική τροπολογία. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε μια υποστήριξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, ξέροντας ότι υπάρχουν διαφορετικές εθνικές εκδοχές για το μοντέλο αυτό. Και το ερώτημα μου τώρα στον εισηγητή είναι το εξής. Το θέμα της εταιρική ευθύνης. Και εδώ είναι το θέμα αν θα πρέπει να παραμείνει αυτό μονάχα στο επίπεδο της εθελοντικής επιλογής. Έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες χρειάζεται να τους ασκηθεί πίεση. Υπάρχουν όμως άλλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πετύχει θαυμάσια πράγματα και μπορούν να είναι ένα υπόδειγμα για τις άλλες επιχειρήσεις. Και εδώ ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα. Είπαμε ότι θέλουμε να τις βοηθήσουμε, αλλά αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μία γιγάντια γραφειοκρατία για να το κάνουμε αυτό, καλύτερα όχι. Εγώ πιστεύω ότι είναι πιο καλό να δίνουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις παρά να προσπαθούμε να τους επιβάλλουμε κάτι. Και από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος υπήρξε ήδη μία η ευρεία υποστήριξη για τις καλές συμβαστικές τροπολογίες που μπορείς να βρεις. Λοιπόν, ας μην μιλάμε για κόλαση, δεν βρισκόμαστε στην κόλαση. Καλώς, μα κύριε Μπαζνά, έχετε ήδη πάρει το λόγο, οπότε... Ξαναμίλησα, το ξέρω, αλλά δύο πράγματα που ήθελα να πω. Ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί το ξέχασα, γιατί κατάφερε να επιτύχει συνένεση σε τόσες πολλές τροπολογίες. Και σκέφτηκα ότι αυτό έπρεπε να το πω το εισηγητή. Το δεύτερο, για τη συμβαστική τροπολογία ε, ΣΥΓΜΑΤΑΦ ταφ, είμαστε ακόμα διαθέσιμοι να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Ωραία. Θέλετε να πάρετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους όσοι πήραν το λόγο. Πολύ χαίρομαι για τόσα άκουσα. Πρόεδρος, καλώς. Μερικές φορές η συζήτηση είναι πράγματι χρήσιμη λοιπόν. Οπότε θα ψηφίσουμε αύριο την έκθεση αυτή. Περάμε στο επόμενο σημείο, σημείο 5 στην ημερήσια διάταξη και θα δώσω το λόγο στην κυρία Σαγιά, δεν είναι εδώ. Alors, Donc, euh, nous avons... Λοιπόν, πράγματι, το σημείο 5 πήγε στο σημείο 9 και το σημείο 9 στο σημείο 5. Οπότε είμαστε στο παλιό σημείο 9 και δίνω το λόγο στην κυρία Λόπε Φοντανιέ για την πέμπτη έκθεση της Επιτροπής όσον αφορά τη συνοχή και τη στρατηγική σχετικά με την πολιτική συνοχής μετά το 2013. Όπως είπαμε, έχουμε προβλήματα επικάλυψης με την Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων. Ελπίζω οι δύο να τα καταφέρουν μεταξύ τους. Αλλιώς θα πάμε στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Έχετε συνεπώς το λόγο κυρία Φοντανιέ, για να μας παρουσιάσετε τη γνωμοδότησή σας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, ήδη μέχρι τώρα είχα διάφορες συναντήσεις με τον εισηγητή από την Περιφερειακή Επιτροπή και ελπίζω ότι τελικά δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα και συνεχίζω στα ισπανικά, λέει η μιλήτρια. Η πολιτική συνοχής όπου περιλαμβάνεται το Κοινωνικό Ευρωπαϊκό Ταμείο, έχει φτάσει στο επίπεδο της πέμπτης ε, έκθεσης για την ε, στρατηγική σχετικά με την πολιτική συνοχή. Συμμετέχει για την καταπολέμηση της ανεργίας και για μια αηφόρο ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική συνοχή πρέπει να εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο, λαμβάνοντας υπόψη πάνω απ' όλα την κατάσταση μέσα στην οποία βρισκόμαστε. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, επειδή ακριβώς έχουμε κρίση και επειδή πλήττονται πολλές οικονομίες μας, διαπιστώνουμε ότι καταστρέφονται συνεχώς επιχειρήσεις και ότι τα επίπεδα ανεργίας έχουν φτάσει σε υπερβολικό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν είναι αναγκαίο να έχουμε μια ισχυρή πολιτική συνοχής με κατάλληλη πρικοδότηση. Η σημερινή κρίση μας έχει δώσει πολλά μαθήματα και ένα από αυτά είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξεπεράσει τις δικές της εσωτερικές ανισορροπίες και να έχει μέλλον. Η πολιτική συνοχής είναι ένα στοιχείο κλειδί για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Στην στρατηγική της Λισαβόνας, που μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει λειτουργήσει, είναι αναγκαίο περισσότερο από ποτέ η στρατηγική 2020 αυτή τη φορά να λειτουργήσει ώστε τα κράτη-μέλη και όλες οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πετύχουν τους στόχους τους. Η πολιτική συνοχής δεν θα αποτελέσει η εξαίρεση και πρέπει να υιοθετηθεί κατά προτεραιότητα με πόρους που θα συνεισφέρουν στην υλοποίησή της. Γι' αυτό ακριβώς είναι αναγκαίο θεματικά να επικεντρωθεί η πολιτική αυτή συνοχή για να μην υπάρξει δεσκοπισμό ε, χρημάτων κονδυλίων σε διάφορε προτεραιότητε. Η θεματική συγκέντρωση που προτείνει η Επιτροπή μα θα δώσει τι κατάλληλε απαντήσει σε συγκεκριμένους στόχους τα επόμενα χρόνια, στόχους που περιλαμβάνονται στη στρατηγική για το 2020. Και για να υπάρξει καλύτερη απόδοση των επενδύσεων πρέπει να φροντίσουμε οι πολιτικές μας να είναι πιο αποτελεσματικές με συγκεκριμένα αποτελέσματα και μάλιστα ποσοτικά εκφρασμένα. Πρέπει να δράσουμε με μεγαλύτερη ευθεία, να φροντίσουμε οι δαπάνες να πηγαίνουν σε συγκεκριμένους τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσφέρουν πρόσθετη αξία σύμφωνα με αυτά που πιστεύουν οι εθνικές, περιφερειακές αλλά και τοπικές αρχές. Χθε στην Περιφερειακή Επιτροπή είπαμε ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την τοπική αυτοδιοίκηση και πιστεύω και εγώ ότι αυτό είναι αναγκαίο για να λειτουργήσουν καλά οι πολιτικές μας. Επίσης πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στα αποτελέσματα. Και γι' αυτό χρειάζεται από πριν να καθορίζουμε σαφείς στόχους και στόχους ποσοτικά εκφρασμένους. Να έχουμε συγκεκριμένους δείκτες και η αξιολόγηση να γίνεται με μεγάλη διαφάνεια. Είναι επίσης αναγκαίο να υπάρχει ελαστικότητα και να μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο το διοικητικό άχθος, το οποίο επομίζονται διάφοροι φορείς που ε, χρησιμοποιούν τα κονδύλια. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει συνεισφέρει κατά πολύ για να μειωθεί ο αντίκτυπος της κρίσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους. Ε, έχει ρόλο κλειδί στην κρίση αυτή. Κρίση η οποία κατέδειξε ακόμα περισσότερο ότι πολιτική συνοχή είναι αναγκαία διότι βοηθάει την αντιγωνιστικότητα των περιφερειών και δημιουργεί θέσει απασχόληση. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να επικεντρώσει τι προσπαθίε του στη δημιουργία απασχόληση και γι' αυτό είναι ζωτική σημασία να υπάρχει διαβίου κατάρτιση ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να προσαρμόσουν τις δεξιοτεχνίες τους στις νέες ανάγκες της αγοράς. Η κρίση επίσης απαιτεί αλλαγές ώστε να έρθουμε και να ενισχύσουμε τους τομείς της νέας οικονομίας που απαιτούν νέες ε, δεξιοτεχνίες και νέα προσόντα. Επίσης πρέπει να διευκολύνουμε τη δημιουργία νέων ε, επιχειρήσεων, διότι αυτές δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να προχωρήσουν με νέα καινοτόμα προγράμματα συνεχίζει στα γαλλικά μιλήτρια. Αυτό είναι το περιεχόμενο της σημερινής μου πρότασης και περιμένω τα σχόλιά σας και τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Σρέτερ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήταν σαφής τώρα η στοχοθεσία από την πλευρά της εισηγήτριας. Εγώ δεν έχω τώρα κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα με το κείμενο αυτό, αλλά πρέπει να υπενθυμίσω ότι είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση που αυτό το κείμενο θα είναι το περιεχόμενο ουσιαστικό της δικής μας συμβολής στη δημιουργία ενός γενικότερου πλαισίου για τα διαφορετικά ταμεία. Επομένως θα πρέπει αυτά τα οποία περιέχονται σε αυτό το έγγραφο να είναι έγκυρα. Ο κύριος Πίπερα από την Περιφερειακή Επιτροπή έχει παρουσιάσει μια έκθεση η οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Τουλάχιστον στην, ε, του, στην αρχική του γλώσσα το κείμενο είναι πολύ καλό. Δυστυχώς δεν είναι τόσο καλή μετάφραση. Επομένως, ανέφερε ότι πρέπει να υπάρχει η συνεργασία του Περιφερειακού Ταμείου με το Κοινωνικό Ταμείο και ότι αυτά είναι απαραίτητα για τις βασικές, το βασικό πλαίσιο της έκθεσης και το περιεχόμενο. Αν δει λοιπόν κανείς την ε, έκθεση Πίπερ, θα πρέπει να καταλάβει πώς θα πρέπει να υπάρχει και η δική μας συμβολή από την Κοινωνική Επιτροπή. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση για όλα αυτά τα πράγματα, αλλά θα πρέπει να καταβάλουμε την προσπάθεια να είμαστε όσο δυνατόν πιο συγκεκριμένοι. Αλλιώς δεν θα το επιτύχουμε ποτέ. Δεν νομίζω ότι αυτό πηγαίνει αντίθετα στις ε, ε, προθέσεις σας, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναλάβουν όλοι οι εισηγητές, οι σκιώδεις εισηγητές και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μας, ώστε να μην χαθούν αυτά τα θέματα από την έχει να κάνει με την καταπολέμηση της ένδυας και τον κοινωνικό αποκλεισμό είναι δικά μας θέματα, θέματα της Επιτροπής μας. Μπορούμε τα θέματα τα οποία διαφορετικά να τα δούμε με τις άλλες επιτροπές, αλλά αυτά τα συγκεκριμένα θέματα είναι δικά μας. Και η Επιτροπή μας όχι μονάχα έχει τα θέματα αυτά στις αρμοδιότητες, αλλά έχει και την γνώση την απαραίτητη για να τα διαλάβει τα θέματα αυτά. Σας λέω και πάλι δεν υπάρχει μία ουσιαστική διαμάχη σε σχέση με το περιεχόμενο, αλλά είναι απαραίτητο να συγκεκριμενοποιηθεί το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου και σε αυτό θα στοχεύσουν οι τροπολογίες μας. Δεύτερο, επί του περιεχομένου και πάλι, εσείς έχετε εστιάσει στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στον χώρο της εργασίας οι οποίοι πρέπει να τύχουν περισσότερη κατάρτισης και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες εργασίας σε μια εποχή κρίσης, σε μια εποχή ε, οικολογικής μεταρρύθμισης και αναπροσανατολισμού της οικονομίας. Ναι, σας υποστηρίζω 100%. Αλλά υπάρχει και ο αγώνας κατά της ε, ένδυας και του αποκλεισμού και έχουμε καταφέρει να έχουμε σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές που ξεφεύγουν από αυτό το στενό πλαίσιο της εργασίας και αντιμετωπίζουν και ανθρώπους που βρίσκονται εκτός αυτού του πλαισίου αποκλειστικά της εργασίας. Είναι ένας από τους στόχους της Ευρώπης 2020 να υποστηρίξει την καταπολέμηση της ένδυας και του αποκλεισμού. Πιστεύω και οι δύο κατευθύνσεις πρέπει να ακολουθηθούν επομένως. Τρίτη παρατήρηση. Πρέπει να υπάρχει και η αρχή της εταιρικότητος, να υπάρχει πραγματικά η συμμετοχή <clears throat> για την ε, από κοινού λήψη απόφασης. Θα πρέπει να διατηρώσουμε λοιπόν τις απαραίτητες ποιότητες που πρέπει να υπάρχουν στο κοινωνικό ταμείο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Επομένως όταν έχουμε μια τέτοια έκθεση η οποία ζητάει συγκεκριμένες μελέτες σε αυτά τα σημεία, εδώ θα πρέπει να έχει μια πραγματική συγκεκριμένη μορφή. Και τελευταία παρατήρηση, η οποία και αυτή είναι σημαντική για μένα, γιατί νομίζω ότι εδώ υπάρχει και μία επικάλυψη με την έκθεση FORM, μάλλον με την, συγγνώμη, με την Επιτροπή Γυναικών, με τι αρμοδιότητε τη επιτροπή Γυναικών. Εδώ είναι απαραίτητο να σκεφτούμε και το ρόλο των γυναικών, να μην τύχαν διακρίσεις, να έχουν ίση αμοιβή για ίση εργασία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έχουμε ζητήσει να υπάρξει μια έκθεση από την Κομισιόν, διότι έχουμε δει ότι σε πάρα πολλά κράτη-μέλη αυτά τα θέματα ισότητα δεν αντιμετωπίζονται σχεδόν καθόλου. Ένα από του στόχου του κοινωνικού ταμείου και τη συνθήκη είναι να γίνει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτό παραγνωρίζεται από πολλά κράτη-μέλη. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει και περαιτέρω προσπάθεια. Ευχαριστώ αγαπητή Αντιπρόεδρε. Αλλά ξέρετε μια γνωμοδότηση πόσο, έστω και σε ενισχυμένη συνεργασία, πόσο μας ε, ε, πιέζει. Ε, καθένα μας ξέρει ότι όταν υπάρχουν παρόμοιες πιέσεις, ε, τι γίνεται. Κύριε Φοντανιέ, τι μας είπατε ξεκινώντας ότι είχατε καλές επαφές με τον κύριο Φάιφερ, Πίπερ, Πίπερ συγγνώμη, αλλά δεν τα αποτελέσματα αυτών των διαβολεύσεων. Τι γίνεται, ο κ. Σπίπερ, θα διαγράψει αυτό το σημείο που έχει να κάνει με την αρμοδική, μοναδική αρμοδιότητα τη Επιτροπή. Εντάξει, δεν είναι μόνο να λέμε ότι τι ωραία, τι καλά, τι ευγενικά, αλλά ο στόχο είναι όλα αυτά να μην ε, συμπεριληφθούν στο μέρο που θα ψηφιστεί από την Επιτροπή την Περιφερειακή. Ναι. Κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι η μας θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Επιτροπής μας, αλλά ναι, με τον κύριο Πίπερ καλή σχέση, καλό άλλο είναι αυτό όμως και άλλο το ότι μετά εμείς θα υποβάλουμε τη δική μας την έκθεση με τα δικά μας τα συμπεράσματα ακριβώς που δεν είναι ότι πρέπει να είναι οπωσδήποτε τα ίδια με τον κύριο Πίπερ, όλα αυτά χρειάζεται να τα συζητήσουμε τώρα προσεχώς. Εντάξει λέει, θα προσπαθήσω όμως να συμβαδίσω όσο γίνεται περισσότερο με αυτά. Το όχι, όχι, όχι για το κοινωνικό ταμείο το ευρωπαϊκό, όχι εδώ είναι εδώ, έτσι για μας. Ε, εντάξει, τελεία και παύλα σε αυτό. Λουισμένοβα και μετά ο κύριος Τσίμερ. Κυρία Τσίμερ, συγγνώμη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε την κυρία Λόπε Φοντανέ να την συγχαρώ σαν σκιώδη συγγήτρια από τους φιλελεύθερους και είναι καλοσυνταγμένο αυτό το κείμενο γνωμοδότησης που συμπεριλαμβάνει πολλά σημεία από εκείνα μας απασχολούν και είναι αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Τα συμπεράσματα και συστάσεις της πέμπτης έκθεσης νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα θέτη ε, σημαντικά τώρα σε αυτή την κρίση την οικονομική και θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά όσο γίνεται καλύτερα για να αποκαταστήσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία και θέση εργασία να δημιουργήσουμε. Βέβαια ε, όλα αυτά δείχνουν και καλή πρόοδο όσον αφορά την ε, ε, συνοχή και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούν να απαλληφθούν οι ανισότητες οικονομικές και κοινωνικές στην Ευρώπη για να δώσουμε τη μάχη μας κατά της φτώχειας και κατά της ανώδης ανεργίας και υποστηρίζω την εισηγήτρια ότι θα πρέπει το συνδυασμό ανάμεσα στο κοινωνικό ταμείο και στο περιφερειακό ταμείο αυτό το συνδυασμό τον κάνουμε καλύτερο όσο γίνεται και ότι θα πρέπει επίσης και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την γεωργική ανάπτυξη να μπορεί να συμμετέχει όπως επίσης και τα οριζόντια προγράμματα Τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης συνδυασμένε προσπάθειες στους κύριους τομείς όπως την ανώσιμη ενέργεια, μόρφωση, κατάρτιση, έρευνα, καινοτομία, όλα αυτά. Με τον τρόπο αυτό και με αυτές τις νορισμένες προσπάθειες, με ένα καλό στόχο για τις κύριες προτεραιότητες. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ασκήσουμε μια πολιτική συνοχή αποτελεσματική και να πετύχουμε τους στόχους της στρατηγικής ε, Ευρώπη 2020 Καταλήγοντας δεν να προσθέσω κάτι ότι θεωρώ τρομερά σημαντικά την ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης και θα πρέπει να καλύψει περισσότερο τις περιφερειακές τοπικές αρχές όπως του και τους εταίρους, τους κοινωνικούς οικονομικούς για να ανταποκριθούμε όσο γίνεται περισσότερο στις προκλήσεις που δημιουργεί αυτή η στρατηγική Ευρώπη 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος. Ευχαριστώ Ε, που σας ευχαριστώ που σας ακούω να μιλάτε στα γαλλικά τη γλώσσα του Ρωσό, του Βολτέρου. Πολύ καλό αυτό. Κυρία Τσίμερ και μετά το Μασμάν. Πάρα πολύ σύντομα από τη δική μου πλευρά. Εγώ θέλω να υποστηρίξω τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί ώστε εμείς να διατηρήσουμε την αρμοδιότητά μας για την ε, μελλοντική διαμόρφωση των ε, δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και για το γεγονός ότι θα πρέπει να έχουμε μια σαφή θέση να της Περιφερειακής Επιτροπής για τα θέματα αυτά. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε φυσικά με την Περιφερειακή Επιτροπή και μέσα στο πολύ περιορισμένο όριο του αριθμού των χαρακτήρων της γνωμοδότησης, σίγουρα εμείς θα πρέπει να παρουσιάσουμε τη θέση μας και αυτό μπορεί να βελτιωθεί και με τις ε, τροπολογίες. Μπορούμε να έχουμε μια κριτική θέση και συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Σρόντερ ότι θα πρέπει εμείς να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις και να υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις στη γνωμοδότησή μας αυτή. Ενώ οι γενικές ε, παρατηρήσεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετούν ακριβώς τον στόχο της ε, κατάδειξης της τάσεω μας. Θα πρέπει να είναι σαφέστερο ποιοι είναι οι δείκτες οι οποίοι θα πρέπει να προταχθούν, προς τα πού θα πρέπει να κατευθυνθούμε, ποια θα πρέπει να είναι η σαφέστερη στοχοθεσία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, πώς θα γίνει ελέγξιμη, πώς θα γίνει με πιο διάφανο τρόπο εφαρμόσιμη και στην πράξη. Και εδώ θέλω να υπενθυμίσω ότι μία από τις ε, διεκδικήσεις μας που προέρχονται από την αλληλεγγύη με τα άτομα τα οποία είναι σε αποκλεισμού και σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού είναι ακριβώς να διευρύνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να αντιμετωπίσει και αυτές τις πτυχές της ε, ε ένδυας και του κοινωνικού αποκλεισμού που μέχρι στιγμής έχουν αντιμετωπιστεί μονάχα με εμβαλ, εμβαλωματικό χαρακτήρα και με ασαφείς διακηρύξεις και εκεί σε αυτό το τομέα πρέπει να πράξουμε κάτι πράγματι. Ο κύριος Τόμας Μαν και μετά η κυρία Edith Power. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Τόμας Μαν και εγώ θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου προς την Βερονίκ για την ευκαιρία που μας έχει δώσει να προχωρήσουμε στη συζήτηση μιας τέτοιας έκθεσης και για τη βάση την οποία έχει παρουσιάσει. Η Βερονίκ έχει σταθεί σε ένα βασικό σημείο στοχοδεσία, ότι πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να είναι ορατότατο και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια σαφέστερη στοχοδεσία. Δεύτερον, Χρειαζόμαστε μια προσέγγιση που έχει σαν στόχο τα αποτελέσματα. Και δεν πρέπει να παρουσιάζεται το κοινωνικό ταμείο ως ένα νεφελώδες ταμείο σε σχέση με, άλλους, με άλλα ταμεία τα οποία έχουν πιο συγκεκριμένους στόχους. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερη εστίαση και καλύτερη στοχοθεσία και σίγουρα ελπίζουμε ότι μαζί με την εισηγήτρια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε σε συγκεκριμένες ε, λεπτομέρειες. Πρέπει το κοινωνικό ταμείο να είναι πιο ορατό στις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολλές από τις πρωτοβουλίες που θέλαμε εμείς να αναπτύξουμε. Η ευκαιρία επίσης να αντιμετωπίσουμε την ε, ένδια και τον κοινωνικό αποκλεισμό ε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι ένας από τους κύριους στόχους μας να πούμε ότι ναι, μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και επομένως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει και μια σαφής οριοθέτηση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού ε, Περιφερειακού Ταμείου. Η εντύπωση που δίνουν μερικές φορές ορισμένα από την Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να πάνε μαζί. Όχι. Εγώ θέλω να εξασφαλίσουμε μια σαφήνεια για το ποιο είναι υπεύθυνο για ποια κατεύθυνση και ποιο πρέπει να είναι ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι με τον κύριο Πίπερ μπορούμε να έχουμε μια καλή συνεργασία. Δεν νομίζω ότι ε, είναι λανθασμένα αυτά τα οποία αναφέρει και εδώ συμφωνώ με την Ελίζαβεθ. Αλλά η Επιτροπή αυτή ε, θα πρέπει θα πρέπει να λειτουργήσουμε βάσει του άρθρου 50 της ενισχυμένης συνεργασίας. Δεν πρόκειται για μια επιτροπή η οποία είναι η αρμόδια της αρχής, και εμείς απλώς γνωμοδοτική. Θα έπρεπε να λειτουργήσει το άρθρο 50 για να έχουμε μια σαφέστερη άποψη για το τι γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ποιοι θα πρέπει να είναι οι στόχοι. Και θέλω να κλείσω με ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει μας πάρα πολύ. Το ποσοστό αυτών που εγκαταλείπουν το σχολείο. Θα πρέπει να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα που θα είναι αποτελεσματικά γιατί πάρα πολλοί δήμοι και πάρα πολλές τοπικές αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν χρήματα για αυτά. Εμείς θέλουμε με τα ευρωπαϊκά χρήματα να δώσουμε τη δυνατότητα τα άτομα αυτά τα οποία φεύγουν από το σχολείο να έχουν κάποια θέση μαθητείας, να έχουν τη δυνατότητα να μπουν και πάλι στο χώρο εργασίας. Και νομίζω ότι το έγγραφο της Βερόνικα είναι ακριβώς η βάση η οποία θα μας επιτρέψει να δώσουμε ένα σαφές μέλλον στο Ευρωπαϊκό και Κοινωνικό Ταμείο και όχι να διαχυθεί σε ένα ασαφή χώρο που περιλαμβάνει και κοινωνικά και περιφερειακά θέματα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή πρέπει να είναι μια έκθεση με την οποία θα αντιμετωπίσουμε τις ε, μέρημνες των πολιτών μας. Θα ήθελα να κάνω μερικά παρατήρησεις, ε, μερικά σχόλια σχετικά με, την, ε, το θέμα αυτό. Όταν ασχολούμεθα με το μέλλον της πολιτικής συνοχής ε, βλέπουμε αρκετά έγγραφα τα οποία παρουσιάζονται, υποβάλλονται και εγώ συντάσω μια γνωμοδότηση που θα έρθει αύριο στα πλαίσια της ημερήσιας διάταξης. Γι' αυτό ακριβώς ε, εκτιμώ, μπορώ να πω, γιατί βλέπω τις πιέσεις που ασκούνται και ότι είναι δύσκολο να τα σεβαστούμε όλα αυτά, όπως είπε και η Βερονίκ. Υπάρχουν επίσης πιέσεις λόγω της ενισχυμένης συνεργασίας και φαίνεται καθαρά άλλωστε ότι το, τα ταμεία λειτουργούν βέβαια ολοκληρωμένα, αλλά και μια μικρή επιχείρηση, ένα όργανο ή κάτι άλλο και υπάρχει ανάγκη για κονδύλια, για τη δημιουργία μας θέσεων απασχόλησης, θα πρέπει να απευθυνθούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Γι' αυτό με σωστό ολοκληρωμένο τρόπο θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα διαθέσιμα κονδύλια. Δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε στο μέλλον τις ε, δραστηριότητε. Δεν μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις ξεχωριστά πάντα. Έτσι και εδώ στην επιτροπή μας στη μια απόφαση και σε άλλη επιτροπή διαφορετική απόφαση γιατί ίσως δημιουργήσει προβλήματα κάτι παρόμοιο. Και ακόμη θα πρέπει να υποβάλουμε σε τροπολογίες για τη συμπλήρωση της έκθεσης για τη στρατηγική του 2020 και προς τα εκεί θα στοχεύσουν αυτή η πόρια, αυτά τα κονδύλια για να δούμε μέχρι ποιο σημείο η στρατηγική αυτή ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ε, πολιτικής συνοχής. Αυτή η πολιτική και η στρατηγική του 2020 εναρμονίζονται, συνδυάζονται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ευρύτερο από τη στατική του 2020 ή μήπως συμβαίνει και το αντίθετο. Το αντίθετο ψιθυρίζει η πρόεδρος, ο κ. Σαρκάς. Και μετά και οι υπόλοιποι, εντάξει. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν συντομία, εν συντομία και αντικαθιστώντας τη σχεδόν ηγήτρια της ομάδας μας που δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα, θα ήθελα να σας μεταφέρω τη συνολική θέση της ομάδας μας, η οποία υποστηρίζει πλήρως την έκθεση της κυρίας Βερόνικα Λόπες Φοντάνια. Νομίζω ότι κάνει μια σαφή διάκριση μεταξύ αυτού που είναι η πολιτική συνοχή, το Ταμείο Συνοχής δηλαδή, και μέσα σε αυτή τη διαδικασία το τι πρέπει να κάνει το κοινωνικό ταμείο. Πρέπει λοιπόν μέσα στη διαδικασία του άρθρου 50 να εξασφαλίσουμε ότι εμείς θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα καθορίσουμε το πώς θα λειτουργήσει το κοινωνικό ταμείο, το οποίο έχει ειδικού στόχους, ειδικέ αρμοδιότητες και είναι ένα κέριο εργαλείο για την κοινωνική ολοκλήρωση. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι στο μέλλον θα υπάρξουν μεγάλες πιέσεις ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να αλλοιωθεί ή να αναμειχθεί με άλλε πολιτικές. Ήδη από τώρα με την έκθεση αυτή εμεί θα πρέπει να είμαστε απόλυτα επάγρυπνοι, να μην ε, βρεθεί υποταγμένη η κοινωνική πολιτική σε άλλες κατευθύνσεις οι οποίες μπορεί να είναι λογικές και αποτελούν τμήμα της πολιτικής συνοχής, αλλά η πολιτική συνοχής δεν μπορεί να καλύψει τις ιδιαιτερότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Επομένω υποστηρίζουμε απόλυτα την Βερονίκ και πρέπει όλοι να αποδεθούμε σε αυτή τη μάχη, όχι μια μάχη με αιματοχυσίες σίγουρα, αλλά μια μάχη ώστε να μην μπει από την κερκόπορτα μια μορφή κυδαιμονίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που, είναι μια πολιτική, που ε, ασκεί μια πολιτική που είναι σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία λέει η πρόοδο. Κυρία Εισηγήτρια, θέλετε να λάβετε και πάλι το λόγο. Ναι, πάρα πολύ σύντομα για να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις και να σας πω ότι έχω απόλυτη επίγνωση των περιορισμών αυτού του κειμένου, ότι είναι ίσως υπερβολικά γενικόλογο, αλλά είναι δύσκολο να είμαστε συγκεκριμένοι και εκπεφρασμένοι με τέτοια τέτοιο περιορισμό όγκου στο κείμενο. Περιμένω από όλε τις πολιτικές ομάδες να βελτιώσουν αυτό το κείμενο και να προσπαθήσουν να συνεισφέρουν όλα αυτά τα σημεία τα οποία μας ενδιαφέρουν ω Επιτροπή απασχόληση και Κοινωνικών Θεμάτων πάντα μέσα στο όριο αυτό των διαβόητων 1500 χαρακτήρων για μια γρομοδότηση. Αλλά σίγουρα εγώ θα έχω την κάθε καλή πρόθεση να φτάσουμε σε ένα θετικό κείμενο. Σας ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος. Επειδή έχουν εκδηλωθεί, η, έχει εκδηλωθεί η διαδήλωση να κατατεθούν τροπολογίες, έχουμε περιθώριο για κατάθεση τροπολογιών που προσδιορίζεται από την ανάγκη να μην, κατα... να μην φτάσουμε καθυστερημένοι στη διαδικασία μεταρρύθμισης των διαφορετικών ταμείων. Επομένως, η εξέταση είναι 17 Μαΐου η προθεσμία για τις τροπολογίες. 24 Μαΐου θα ξεκινήσει η εξέταση των τροπολογιών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κατατεθούν στα αγγλικά ή στα γαλλικά. 19 Απριλίου. 19 Απριλίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες και 24 ε, Μαΐου είναι η συζήτηση στην Επιτροπή μας. Το πρωί 24 Μαρτίου, απόγευμα 24 Μαΐου θα γίνει η ψηφοφορία και 26 Μαΐου θα αποφανθεί η Περιφερειακή Επιτροπή. Ελπίζουμε ότι μέχρι τότε θα έχουμε επιλύσει όλα τα προβλήματα αυτά της επικάλυψης των αρμοδιοτήτων. Σημείο 6 τώρα της της διάταξης και συγκεκριμένα γνωμοδότηση της κυρίας Jean Λαμπέρ για τη χρήση των ραδιενεργών αποβλήτων και των εξυντλημένων καυσίμων Υπάρχουν κάποιε τροπολογίε οι οποίες θεωρήθησαν μη παραδεκτές γιατί εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων επιτροπών και όχι της ειδική μας. Και αυτή η θέση καταλήξαμε σε αυτή τη θέση με τη συμφωνία όλων των εμπλεκομένων πολιτικών ομάδων. Σας δίνω το λόγο λοιπόν κυρία εισηγήτρια για να παρουσιάσετε τις συμβαστικά τροπολογίες που έχουν αναλωθεί επί της εκθέσεώς σας. Η κυρία Κορνέλης ε, την κυρία Τζιν Λάμπερτ. Ναι, η Τζιν δεν μπορούσε να έρθει εδώ και μου είπε μου ζήτησε να την ε, εκπροσωπήσω. Θα ήθελε η συγγήτρια να ευχαριστήσει όλου του σκιώδει εισηγητέ για την τόσο θετική συνεργασία του και τι πάρα πολύ χρήσιμε ανταλλαγέ απόψεων. Ζητά συγγνώμη για το γεγονό ότι δεν μπορεί να είναι σωματικά παρούσα στην τρέχουσα συνεδρίαση. Παρά το γεγονό ότι τα τρέχοντα γεγονότα στην Ιαπωνία έχουν θέσει ένα αμφιβόλο το θέμα τη ασφάλεια τη πυρηνική ενέργεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι το σχέδιο γνωμοδότηση και τροπολογία έχουν πριν από την καταστροφή τη Φουκουσίμα. Ο στόχο τη είναι όχι να αντιμετωπίσει το θέμα της ποινική ενέργειας εν γέννη, αλλά να εστιάσει στα θέματα υγείας και ασφάλειας όλων των εργαζομένων. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους σκιώδεις εισηγητές για την υποστήριξη αυτής της γενικής κατεύθυνσης της κυρίας εισηγητής. Έγιναν συμβαστικές τροπολογίες για το άρθρο 9, για την εμπειρογνωμοσύνη και τις ε, ε, επιδεξιότητες και επίσης για το άρθρο 12 για την διαφάνεια και επίσης μια τροπολογία για το χρονικό πλαίσιο. Άρθρο 4 προσπάθησε η εισηγήτρια να έχει την μεγαλύτερη δυνατή συνένεση και ενσωμάτωσε τις προτάσεις των πολιτικών ομάδων στις προτάσεις της. Κάποιες προφορικές τροπολογίες επροτάθησαν επίση σε σχέση με την συμφωνία των σκιωδών εισηγητών στην αρχή της εβδομάδας. Σας ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας για την υποστήριξή σας, ιδίως για τη διεύρυνση της εμβελίας αυτής της ε, οδηγίας που να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που μπορούν να, έχουν, να κάνουν συνεργασία τους με τα αναλωμένα καύσιμα και τα απόβλητα, τα διενεργά, και επίσης για την αλλαγή της νομικής βάσης που μπορεί να τους καλύψει και για όλους τους άλλους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από τη διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων και αναλωμένων καυσίμων και προσβλέπω στα σχολεία σας. Μερσή. Ευχαριστώ πολύ λέει η κυρία Φιγκυρέντου. Έχουμε εδώ δύο ομιλητές που έχουν, ε, έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Μάισνερ. Σας, έδαμε. Ε, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω, αντίθετα από αυτό που κάναμε τον κύριο Φάλμπουρ, που το ξέχασα, να πω ευχαριστώ από την αρχή στην εισηγήτρια και αυτή βέβαια είναι ιδιαίτερα επίκαιρη η γνωμοδότηση, όπως είπε και η κυρία Κορνέλσον, μετά από τα γεγονότα της Φούκου Σήμα. Αλλά έχει ένα γενικό χαρακτήρα, πρόκειται μια γενική ρύθμιση. Τώρα βέβαια μπορούμε να δούμε τα θέματα αυτά λίγο πιο ενδελεχώς. Τα θέματα της προστασίας και της, της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα αυτό. Εγώ βρίσκω ότι είναι μια πολύ καλή έκθεση, μια καλή γνωμοδότηση συγκεκριμένα. Και επίσης νομίζω ότι με τις συμβαστικές τροπολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 ότι υπάρχει μια πολύ καλύτερη διατύπωση. Γιατί είχαμε πει ότι πρέπει να υπάρχει ασφάλεια για 150 χρόνια, η ασφάλεια για 250 χρόνια, τώρα είναι πολύ καλύτερη η διατύπωση όσο είναι επιβλαβή για τους εργαζόμενους και το περιβάλλον αυτά τα απόβλητα. Αυτή είναι μια πιο ευτυχής ε, διατύπωση. Επίσης στο σημείο 28 επίση η τροπολογία που κατατέθηκε νομίζω ότι μπορεί να είναι πολυθετική και την υποστηρίζουμε. Δύο ακόμα σημεία θέλω να αναφέρω πρώτα απ' όλα. Για την κυρία Λάμπερτ έχω κάποια προβλήματα με την τροπολογία 21 με την έννοια της γενικής ευθύνης, της γενικής αστικής ευθύνης. Δεν ξέρω πόσο θα μπορούσα να δεχτώ την αντιμετώπιση και επίσης και για την τροπολογία 29 είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν αυτά τα απαραίτητα ανθρώπινα και οικονομικά μέσα για να αντιμετωπιστούν τα απόβλητα αυτά όταν φτάνουν στο τέλος της επικοινωνότητας, είτε είναι 150 ή 250 χρόνια. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο και εγώ θα καταψηφίσω στην τωρινή μορφή τροπολογία 29 γιατί δεν νομίζω ότι είναι εφικτό αυτό το οποίο αναφέρεται στην τροπολογία αυτή. Και επίσης η τροπολογία 80%. που αφορά την αποθήκευση των αποβλήτων μόνο στο κράτος μέλος όπου έχουν προκύψει, όπου έχουν παραχθεί. Βέβαια μπορούμε να έχουμε την αρχή ότι ο Ριπένον πληρώνει, αυτό είναι λογικό. Αλλά οι γεωλογικές δυνατότητες των κρατών μελών για την αποθήκευση αυτών των αποβλήτων είναι πολύ διαφορετικές. Και αν έχουμε στο μέλλον ένα ασφαλές τόπο εναπόθευσης, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, που είναι σε ένα άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο γίνεται η παραγωγή των πυρηνικών αποβλήτων, νομίζω ότι σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πούμε ότι και αυτό, αυτός ο ασφαλής τόπος εναπόθεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί, γιατί για μένα το ουσιαστικό είναι να υπάρξει η ασφαλής εναπόθεση αυτών των αποβλήτων. Γι' αυτό δεν μπορώ να δεχτώ την τροπολογία 81 ή 82 έχει ένα άλλο χαρακτήρα αν μιλάει για τρίτες χώρες, αν είχαμε παραγωγικά μια συμφωνία με την ε, Ρωσία για να αποθηκεύσουμε εκεί ε, απόβλητα, αυτό είναι μια διαφορετική αντιμετώπιση. Θα είχαμε ένα πρόβλημα έτσι και γι' αυτό έχει λογική να πούμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει αναπόθεση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύουμε ότι αυτό δεν πρέπει να καλυφθεί μέσα από τη συνθήκη Ευρατόμ. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα συναπόφαση του Κοινοβουλίου με τη νέα συνθήκη τη Λισαβόνα και το πρόβλημα αυτό έχει έρθει και πάλι στην επικαιρότητα με την Φουκου Σήμα. Σα ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Η κυρία Στάινρουκ έχει το λόγο τώρα. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια η οποία έχει παρουσιάσει μια πολύ πλήρη έκθεση, αλλά επίση θέλω να ευχαριστήσω και την πρόοδο της Επιτροπής μας, η οποία μας ανάφερε χθε για τις ε, τροπολογίες αυτές. Και νομίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό και με την ε, συνεργασία μεταξύ των σχεδιοδών συγκεκριτών έχουμε προχωρήσει ένα βήμα περισσότερο. Και έχουμε καταθέσει, έχουν κατατεθεί και μια σειρά τροπολογίες στην Επιτροπή Βιομηχανίας, οι οποία ήταν αντικείμενο αυτής τη διαβούλευση. Εγώ από την πλευρά της πολιτικής μου ομάδας υποστηρίζω την έκθεση αυτή και τις συμβασικές τροπολογίες, γιατί εδώ θα πρέπει να προταχθεί το γενικό συμφέρον, που είναι ότι η απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η προστασία των εργαζομένων και αυτό θα πρέπει να γίνει και για ένα διάστημα το οποίο θα κρατήσει πολύ καιρό και δεν μπορούμε να προβλέψουμε από σήμερα ακόμα πόσο θα κρατήσει αυτό το διάστημα. Και επίσης το θέμα της αστικής ευθύνης θα πρέπει αυτοί οι οποίοι παράγουν τα απόβλητα να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη χωρίς κανένα περιορισμό. Η έκθεση Λάμπερτ είναι μια πολύ καλή βάση ώστε στα κράτη-μέλη να υπάρξει σωστή αντιμετώπιση της προστασίας των εργαζομένων σε ε, περιοχές που έρχονται σε επαφή με αυτά τα επικίνδυνα απόβλητα και τα κράτη δεν θα πρέπει να είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να αναλάβουν το κόστος όλων αυτών των ενεργειών, αλλά θα πρέπει να εγγυηθούν όταν αυτό είναι απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή θέση στην αυριανή ψηφοφορία που θα τονίσει τη στεναρή θέση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η πρόεδρο. Πρώτου δώσω τον λόγο τώρα στου δύο επόμενου ομιλητέ. Θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση για αυτό το οποίο είπε ήδη στην αρχή τη συνεδρίαση η κυρία Μπερέσου ότι υπήρξε ένα σύνολο τροπολογιών που δεν έγιναν παραδεκτές, γιατί αντιμετωπίζουν θέματα τα οποία εκφεύγουν τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Είναι οι τροπολογίες 5, 15, 16, 52, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 81 αλλά και 82. Δεν θεωρήθηκαν λοιπόν παραδεκτές αυτές οι τροπολογίες γιατί δεν αντιμετωπίζουν θέματα της αρμοδιότητας της δικής μας Επιτροπής και θα πρέπει να λάβετε υπόψη αυτά τα στοιχεία. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους ε, άλλους σκιώδεις εισηγητές. Ο κύριος Τόμας. Ο κύριος Τόμας Μάνι. Τόμας Χέντελ. Είναι μια εξαιρετική εργασία υπό την ε, ηγεσία της κυρίας ε, Λέμπερτ και εμείς έχουμε υποστηρίξει πλήρως την έκθεση αυτή και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό να αγωνιστούμε για τη διεύνηση της νομικής βάσης αυτής της έκθεσης ώστε να υπάρξει μια μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή να έχουμε μια αναφορά για εργασιακά θέματα και τις ε, οδηγίες οι οποίες αφορούν αυτά τα θέματα ήδη. Αυτό είναι πολύ σωστό. Τρίτον, στο κείμενο αυτό το οποίο θα πρέπει να ψηφιστεί αύριο, υπάρχει και η διεύρυνση της εμβέλειας για εργαζόμενους οι οποίοι δεν εργάζονται σε σταθερές, σταθερά με αυτά τα προϊόντα, τα ραδιεργά, αλλά και σε να πελάβει δηλαδή και άτομα τα οποία μπορεί να χρειαστεί να έρθουν σε επαφή με ραδιεργά προϊόντα. Αυτό είναι πολύ σωστό. Ένα ακόμα σημείο το οποίο θέλω να παρουσιάσω και θέλω εδώ την υποστήριξή σας για μια τροπολογία που έχω καταθέσει εγώ ίδιος, στην τροπολογία 90. Από τη δική μου εμπειρία στις ε, συμβάσεις που έχουν να κάνουν με την προστασία από επαγγελματικές ασθένειες και τις ε, επαγγελματικές συντάξεις αναπηρίας ή ασθένειες, νομίζω ότι θα πρέπει να διευρύνουμε την ε, δυνατότητα απόδειξης της μόλυνσης από ραδιενεργά απόβλητα πολλές φορές είναι κάτι στην νομική πρακτική. Είναι πολύ δύσκολο να αποδείξει κανείς ότι έχει λάβει χώρα μία, α, μία μόλυνση με ραδιενεργά υλικά, ακόμα και αν έχει εργαστεί κανείς πολλά χρόνια με αυτά τα υλικά. Γι' αυτό ζητώ στην τροπολογία 90 να κρατώνται τα έγγραφα εργασίας για 50 χρόνια και να, κρατούνται από μια ανεξάρτητη αρχή ώστε με τον τρόπο αυτό να έχουν τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι ακόμα και εκ των υστέρων να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Τόμας Μαν επιτέλους. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και για μένα είναι μια πολύ καλή βάση για να προχωρήσουμε και αυτό βέβαια είναι διαφορετικό θέμα από αυτό το οποίο συζητούσαμε στο Στασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα, το θέμα της γενικότερης ατομικής πολιτικής για την πυρηνική ενέργεια και του θέματος να έχουμε κάποια ε, κατεύθυνση μέσα στο χρόνο. Εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο μας ενδιαφέρει να λάβουμε υπόψη την ασφάλεια των εργαζομένων ξέρουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να έχουμε μια κοινή θέση για την πυρηνική ενέργεια, γιατί έχουμε διαφορετικές θέσεις και διαφορετικές εμπειρίες για την πυρηνική ενέργεια στα κράτη-μέλη και γι' αυτό δεν υπήρξε ένα κοινό ψήφισμα. Αλλά δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. <clears throat> δεν είναι αξιοζήλευτη η θέση του κυρίου Έτιγκερ, ο οποίο προσπαθεί να επιτύχει μια κοινή θέση όταν υπάρχουν τόσε διαφορετικέ απόψει για τα θέματα αυτά. Αλλά αυτό το οποίο έχουμε εδώ στην Επιτροπή μας είναι διαφορετικό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι οποίοι εργάζονται ε, θα πρέπει να προστατευτούν. Δεν θα πρέπει αυτό να εξαρτάται από το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει πυρηνική ενέργεια σε μια χώρα και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν οι παράγοντες ασφάλειας στην εργασία των ανθρώπων αυτών. Ακόμα και αν η ελπίδα μας ήταν να υπάρχει μια γενικότερη κάλυψη για τα θέματα αυτά. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι τα άτομα αυτά όχι μόνο να μπορούν να επιβιώνουν όταν εργάζονται και αντιμετωπίζουν ατυχήματα, αλλά να έχουν μια εγγύηση ότι θα υπάρχει προστασία της υγείας τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να αντιμετωπίσουμε την αστική ευθύνη έναντι των εργαζομένων με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι ευρύς και να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι επαρκής οι διασφαλίσεις. Γιατί ποιος θα πίστευε ότι η Ιαπωνία θα βρισκόταν στην κατάσταση που βρέθηκε σήμερα. Θεωρούσαμε ότι τα εργοστάσια της ήταν ε, ασφαλή. Και ποιος μπορεί ακόμα και στη δική μας χώρα κύριε Χέντελ να δώσει μια απόλυτη εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει ποτέ ένα τέτοιο πρόβλημα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν πέραν αυτό που εργάζονται στα πυρηνικά εργοστάσια, τους μεταφορείς, τις αστυνομικές αρχές, τους πυροσβέστες, όλους αυτούς που είδατε στην Ιαπωνία ότι ακόμα και θελοντικά βρέθηκαν στο εργαστήριο της Φουκουσίμα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ασφάλειά τους και η υγεία τους θα τύχουν προστασίας. Και υπάρχει επίσης και η κατάσταση των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μεταφερθεί σε περιοχές οι οποίες θεωρήθηκαν αρχικά ότι ήταν ασφαλείς ενώ μπορεί να μην είναι. Δεν πρέπει λοιπόν να παραγνωρίσουμε την κατάσταση όλων αυτών των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε έγγραφα τα οποία θα είναι διαθέσιμα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να μπορέσουμε μετά σε, ακόμα και μετά από πολλά χρόνια να κατανοήσουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν διαπράξει λάθη ή έχουν κάνει ενέργειες οι οποίες δεν ήταν επαρκείς. Και αυτό θα είναι ένα θετικό, ε, <clears throat> ένα θετικό μήνυμα για τις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων που χρειάστηκε να μεταφερθούν σε άλλες περιοχές μακριά από τη Φουκουσίμα, να τονίσουμε ότι, υπάρχει, ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι προδιαγραφές για να ελέγχουμε την κατάσταση της υγείας και να προστατεύουμε αυτούς τους ανθρώπους εργαζομένους. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Προεδρεύουσα. Δεν ξέρω αν η κυρία Κονέλσεν θέλει να επανέλθει και να κάνει κάποιο σχόλιο για αυτά τα οποία λέχθηκαν. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Θα μεταφέρω όλα τα συγχαρητήριά σας στην κυρία Λάμπερτς. Και σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Για την κυρία Μάισνερ πρώτα. Όπως και η κυρία Φιγερέδο και η κυρία Στάνκο είπαν, οι δύο τροπολογίες με τις οποίες έχετε πρόβλημα έτσι κι αλλιώς δεν θεωρούνται αποδεκτές, οπότε δεν υπάρχει πια πρόβλημα. Α, εγώ τα μπέρδευσα με αυτό που είπε βοηθό μου και νόμιζα ότι έπρεπε να ψηφίσουμε πάνω σε αυτέ, αλλά τελικά όχι τόσο το καλύτερο. Για την 21, ναι, πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ σημαντική. Έχει να κάνει με την ευθύνη και σημαίνει ότι φροντίζουμε κάποιος να είναι υπεύθυνο και για την υπερεργολαβία, υπερ, υπερ, υπερ Πάντα δηλαδή να υπάρχει κάποιος υπεύθυνο. Ελπίζω να την στηρίξετε την 21 λοιπόν. Κύριε Χάντελ. Αναφερθήκατε στην τροπολογία 90. Η συγκήτρια υποστηρίζει όλες τις τροπολογίες των άλλων πολιτικών ομάδων, έτσι κι αλλιώς. 19 τροπολογίες, συγγνώμη, 19. Νομίζω ότι η μεγάλη μάχη δίνεται μετά. Εκεί πρέπει να, κάνουμε, να δώσουμε αγώνα με τους συναδέρφους από την Ήτρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λοιπόν αύριο θα γίνει η ψηφοφορία αυτής της νομοδότησης. και πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος των προτάσεων που έχουν διατυπωθεί θα μπορέσουν να εγκριθούν. Έτσι έχουμε κλείσει το σημείο αυτό της ημερησίας διατάξεως και περάσαμε στο επόμενο. Η ακρόαση με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε σχέση με την υλοποίηση και την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 94-2008 περί προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση κανονίου ή αφαιρεγιότητας του εργοδότη. Η συγγήτριά μας είναι η κυρία ε, Ουγγέρνε, η κυρια ε η οποια θα παρουσιάσει το θέμα αυτό. Πού είναι? Θα σας δώσω λοιπόν το λόγο αμέσως. αλλά θα περάσουμε στον ούπο στους καλεσμένους μας. Θέλετε το λόγο προηγουμένως ή όχι. Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Περίμενα τη μετάφραση, γι' αυτό άργησα να αντιδράσω. Ευχαριστώ. Τίποτα άλλο. Αλλά τώρα νομίζω ότι καταλάβατε τι είπα. Θέλετε να κάνετε μια παρουσίαση εισαγωγική του θέματος. Εάν ναι, σας δίνω το λόγο. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Αλλά για πείτε μας, πού είναι η κοινωνική εταίρη, πού βρίσκονται εδώ στην αίθουσα για να έχω υπόψη μου, για να ξέρω σε ποιον απευθύνομαι δηλαδή. Εισαγωγικά. Η ρύθμιση αυτή για την ευκαιρεότητα ξεκίνησε τον Μάιο του 2002. Αφορά όλες τις χώρες, έχει να κάνει με όλες τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την πτώχευση, εκτός εάν πρόκειται για ασφάλεια πιστοτικά ιδρύματα. Είναι δηλαδή ένας περιορισμός αυτός. Υπήρχε ένα παλαιότερο καθεστώς που αντικαθιστάται για τη δίκηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει επιπτώσεις και στις διασυνοριακέ περιοχές. Δεν μιλάμε για εναρμόνιση των κανόνων. Ισχύει αυτό και στην Επιτροπή Τζούρι, αν δείτε τη δικιά της έκθεση. Πάντως αλλαγές πρέπει να στηρίζουν τις επιχειρήσεις που δρούν διασυνοριακά και να τις βοηθούν. Να γίνονται επιστροφές στους πιστωτές και να υπάρχει όσο γίνεται μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων. Το 2008 είχαμε μια οδηγία για την προστασία των ε, εργαζομένων από τους εργοδότες. Κάτι διαφορετικό από τη ρύθμιση του 2002. Το σχέδιο έκθεσης πάντως που έχετε μπροστά σας ε, ουσιαστικά είναι η αντίδρασή μας στην Επιτροπή Τζούρι που θέλει να προχωρήσει περισσότερο στο θέμα. Εγώ προσπάθησα στην ε, γνωμοδότησή μου να δω πού χρειάζονται ε, προσαρμογές ή που είναι επιθυμητές οι αλλαγές ή κατά πόσο τα πράγματα λειτουργούν ικανοποιητικά. Γι' αυτό και οργανώσαμε την ακρόαση αυτή, για να ακούσουμε τις επιθυμίες των κοινωνικών εταίρων, τους οποίους καλωσορίζω θερμά εδώ και περιμένω να ακούσω τι έχουν να μας πούνε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η Πρόεδρος. Η γραμματεία μας, λοιπόν, έχει προσκαλέσει τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσία μόνο του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων και στη συνέχεια θα έχουμε μαζί μας και εκπροσώπους από την Κομισιόν. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω δίνον τον λόγο τις, τους εκπροσώπους της, της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας ε, Εργαζομένων, την κυρία Βιν Βάρνικ. Έχετε το λόγο λοιπόν παρακαλώ και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Βάντερμπεργκ. Τα λέω σωστά. Είσαστε οι δυο σας που θα παρέμβετε για αυτό το θέμα. Έτσι δεν είναι. Έχετε το λόγο λοιπόν. Παρακαλώ κύριε Βάνη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που προσκαλέσατε εδώ τους κοινωνικούς εταίρους στην ακρόασή σας. Βέβαια, έχετε τη μία πλευρά των κοινωνικών εταίρων, μόνο τα συνδικάτα έδραξαν την ευκαιρία αυτή και παρευρίσκονται. Σας ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων θεωρεί την οδηγία αυτή για την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση που υπάρχει αφαιρεγκαιότητα του εργοδότη κάτι αναγκαίο για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Προσφέρει την ελάχιστη προστασία στους εργαζόμενους παντού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης είναι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία από τις πιο σημαντικές σήμερα που βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση. Ο κίνδυνος ε, επιχειρήσεις να μην μπορούν να φέρουν σε πέρα τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους εργαζομένους τους, ε, ο αριθμός των επιχειρήσεων αυτών αυξάνει συνεχώς. Και βλέπουμε από το 2008 μέχρι το 2009 είχαμε μια αύξηση της τάξης του 19% περιπτώσεων ε, τόχευσης επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 61% δηλαδή αύξηση όσον αφορά τους εργαζομένους που επηρεάζονται από την πτώχευση αυτή. Η καλύτερη προστασία των εργαζομένων είναι βέβαια να αποφεύγεται η πτώχευση της επιχείρησης στην οποία εργάζονται. Και έτσι έρχομαι στα στοιχεία κλειδί που εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων. Όσον αφορά την οδηγία αυτή για μας, το στοιχείο κλειδί βέβαια είναι το άρθρο 3.1 που αναφέρεται στην προστασία των εργαζομένων και τους ε, ισχυρισμούς που μπορούν να προβάλλουν για πληρωμή. Υπάρχει εθνική νομοθεσία βέβαια σε πάρα πολλές χώρες. Υπάρχουν λοιπόν αυτές, αυτοί οι ισχυρισμοί που πρέπει όμως να διευκρινιστούν περισσότερο. Γιατί πολλές χώρες μέλη έχουν έναν περιοριστικό ορισμό της αμοιβή για παράδειγμα αποκλείουν τα μπόνους, κάποιους διακανονισμούς, επιδόματα κτλ. Εμείς πάντως πιστεύουμε ότι θα έπρεπε αν μη τι άλλο να αφαιρέσουμε το κομμάτι εκείνο το οποίο αναφέρει έτσι όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία ώστε να συμπεριλαμβάνονται και αυτές οι περιπτώσεις και να υπάρχει ένας ευρύς ορισμός του τι χρωστά εργοδότες τους ένα άλλο σημείο που για μας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι το σημείο 4 που αναφέρεται στον περιορισμό της ευθύνη των εγγυητικών οργανισμών. Εδώ έχουμε δύο στοιχεία τα οποία θέλουμε να αναφέρουμε. Το ένα έχει να κάνει με την περίοδο ε, μέσα στην οποία πρέπει να πληρώσει ο εργοδότης και δεύτερον την οροφή, το ανώτατο δηλαδή όριο της πληρωμής. Για μας και τα δύο αυτά σημεία είναι αλληλένδετα μεταξύ τους, γιατί το όριο μπορεί να κριθεί ικανοποιητικό, αλλά αν συνδέεται με ένα πιο μικρό χρονικό διάστημα, ε, θέτει σε κίνδυνο τους ίδιους τους κοινωνικούς στόχους της οδηγίας. Στην πράξη. Αυτό που αναφέρουν πολλά ε, συνδικάτα από την εμπειρία του σε εθνικό επίπεδο είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις μένουν απλήρωτοι οι μισθοί και ξεπερνούν τα όρια που βάζει η εθνική νομοθεσία. Για παράδειγμα στη Γερμανία, αλλά όχι μόνο. Δεν διαφέρει δεν ε, έρχεται ουρανοκατέβατη. Υπάρχουν προηγουμένως ε, προβλήματα ε, οικονομικά του εργοδότη, ο οποίος δεν πληρώνει σε τακτική βάση τους εργαζόμενους. Καθυστερεί τους μισθούς. Η ελάχιστη περίοδος στο άρθρο 4.2 πρέπει να είναι πιο μεγάλη. Και στο άρθρο 4.3 πρέπει να επαναδιατυπώσουμε το κείμενο. Γιατί τι σημαίνει ε, κοινωνικά συμβατό. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη νομική σαφήνεια λοιπόν και να μην περιοριστούν οι υποχρεώσεις των κρατών μελών. Έπειτα πιο συγκεκριμένα, για να έρθουμε στο σχέδιο γνωμοδότησης όσον αφορά το εταιρικό δίκαιο για την αφαιρεγγιότητα. Η ρύθμιση για την αφαιρεγκαιότητα επηρεάζει πάρα πολύ την κατάσταση της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε, οι επιχειρήσεις μπορώ να φανταστώ να επιλέγουν την έδρα τους όχι ανάλογα με τις διαδικασίες αφαιρεγκαιότητας αλλά βάσει άλλων παραγόντων που εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις τους. Φορολόγηση, για παράδειγμα. Εταιρικότητα, επιχειρήσεστε μάλλον τι σημαίνει. Σημαίνει, άμα φτιάχνεις μια επιχείρηση, δεν σκέφτεσαι αμέσως τη δυνατότητα πτώχευσης της επιχείρησής σου. Γι' αυτό και μας εξέπληξε που δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα των νόμων για την απασχόληση και της οδηγίας για την αφαιρεγκαιότητα. ξεκινήσαμε από το 2004. Ο στόχος παραμένει. Είναι ο ίδιος, είναι η προστασία των εργαζόμενων. Η Συνομοσπονδία μας πιστεύει ότι ο στόχος διασφάλισης της ελάχιστης ε, προστασίας καλύπτεται από τη ρύθμιση αυτή. Παρ' όλα αυτά υπάρχει περιθώριο για βελτιώσεις. Οι ισχυρισμοί αποσημείωσης, ε, το χρονικό διάστημα και η οροφή. Πιστεύουμε ότι υπάρχει τεράστια ευελιξία ακόμα για τα κράτη-μέλη. Αναρωτιόμαστε λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα να προσθέσουμε και το θέμα της σωστής ενσωμάτωσης στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας αυτής. Ήδη από τον Φεβρουάριο ξέρουμε ότι γίνονται ε, παραβιάσεις στην κοινοτική νομοθεσία εξαιτία ακριβώ αυτή τη έλλειψη ελέγχου τη ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία. Μήπω λοιπόν θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω η Επιτροπή με προσφυγές υπεραβάση για παράδειγμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Και τώρα για να συμπληρώσει τα λεγόμενά σα, ο κύριο Βαντενμπέργκ έχει το λόγο. Έχετε το λόγο. Και εσείς είσαστε από την Ευρωπαϊκή Νομοσπονδία Συνδικάτων, έτσι δεν είναι είστε οι μόνοι κοινωνικοί εταίροι οι οποίοι δέχτηκαν να συμμετάσχουν σε αυτήν την ακρόαση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριος Φαντενμπέρκ και εγώ θέλω να υποστηρίξω τα σχόλια της συναδέλφου μου και θέλω να σταθώ λιγάκι σε πιο πρακτικά θέματα εφαρμογής για την οδηγία 2008 κάθετος 94 στο Βέλγιο για να καταδείξω τι είναι τα θετικά και τι είναι τα αρνητικά και τα παραθυράκια που έχει αυτή η οδηγία. Γενικά, <clears throat> στο Βέλιο, η κοινωνική εταίροι και τα συνδικάτα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τον τρόπο που έχει εφαρμοστεί αυτή η οδηγία στο Βέλιο πάντα. Και αυτό καταδεικνύεται από το γεγονός ότι έχουμε μια κυβέρνηση χωρίς ουσιαστικές εξουσίες εδώ και σχεδόν ένα χρόνο και παρόλα αυτά καταβάλλονται ακόμα οι αποδοχές των εργαζομένων στο Βέλιο. Υποστηρίζουμε όμως αυτή την οδηγία διότι θεωρούμε ότι η εφαρμογή της δεν έχει τύχη κατάχρησης στην περίπτωση των, για τα παραθυράκια τα οποία υπάρχουν και αυτός είναι ένας λόγος για να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία που έχουμε συγκεντρώσει για να κλείσουμε ορισμένα παραθυράκια στην οδηγία. Για παράδειγμα, <clears throat> βάσει του άρθρου 3 υπάρχουν διεκδικήσεις που περιλαμβάνουν οροφές και περιόδους αναφοράς. Στο παρελθόν ήταν πολύπλοκο το σύστημα με διαφορετικές περιόδους αναφοράς και διαφορετικά, διαφορετικές οροφές σε σχέση με το αν οι διεκδικήσεις αφορούσαν ε, επιδόματα διακοπών ή αμοιβέ, βασικό μισθό ή άλλες πληρωμές. Εμείς απλοποίησαμε το σύστημα στο Βέλγιο Υπάρχει τώρα μια συνολική μονάχα οροφή 25.000 ευρώ, ώστε όλες οι διεκδικήσεις, όλες οι, δια, οι αγωγές αυτές για ποσά κάτω από 25.000 καλύπτονται από το λεγόμενο Fond de Fermeture, το ταμείο που επεμβαίνει όταν κλείσει μια επιχείρηση. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως ατόμων που είχαν πάρει παραγωγός χάρη το επίδομα ε, διακοπών αλλά όχι το πιστό τους και επομένως είχαν, λιγότερα, είχαν πάρει λιγότερα χρήματα από άλλους που πήραν ένα τμήμα του μισθού τους και, το επίδομα, και τα επιδόματά τους. Λοιπόν, για τον πληθυσμό λοιπόν θα ήταν καλύτερο να έχουμε ένα απλό σύστημα και εύληπτο σύστημα. 95% των ε, ποσών που διεκδικούν οι εργαζόμενοι καλύπτεται από ένα φορέα εγγύσεων και σε 80% πληρώνεται το 100% της διεκδίκησης. Και παρόλα αυτά, άμα δείτε τις συνεισφορές με τις οποίες συν, ε, <clears throat> συντηρείται το σύστημα, οι συνεισφορές των εργοδοτών είναι χαμηλότερες από 0,02 του ακαθάριστου, των ακαθαρίστων αποδοχών των εργαζομένων. Δεν είναι λοιπόν ασήμαντο ποσό, αλλά δεν είναι υπέρογκο ποσό, δεν είναι ένα βάρος για τους ε, ε, εργοδότης και θα, που θα τους υποχρέουν να δεν κατασταθούν κάπου αλλού. Και σε ό,τι αφορά την, ε, τον αποκλεισμό ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων, <clears throat> πιστεύω ότι και εδώ υπάρχει σωστή εφαρμογή της οδηγίας στο Βέλιο. Στο παρελθόν οι εργαζόμενοι σε τομείς ε, που εργάζονται σε μη κερδοσκοπικές ε, επιχειρήσεις εξαιρούνται τις εφαρμογή αυτής της οδηγίας, αλλά αυτό έχει αλλάξει από το 2008 όταν ε, υπήρξε μια χρεοκοπία ενός ε, ασύλου για ηλικιωμένους και στην περίπτωση αυτή καλύφθησαν, έπρεπε να καλυφθούν και οι εργαζόμενοι εκεί. Παραμένει ακόμα ο κίνδυνος για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις οι οποίες μπορεί να περάσουν σε αφαιρεγγιότητα. Φυσικά είναι μικρότερο ο κίνδυνο αυτό από ό,τι στι εμπορικέ επιχειρήσει και στην περίπτωση αυτή υπάρχει μια μικρότερη συμβολή που γίνεται για του ε, ε, εργοδότε τέτοιων μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων. Επομένω υπάρχει μια μεγαλύτερη ευκαμψία για να αντιμετωπιστούν οι διάφορε κατηγορίε εργαζομένων. Μια τελευταία παρατήρηση αφορά τις διαμεθοριακές και διακρατικές καταστάσεις και προβλήματα. Εδώ στο Βέλγιο το Fond de Fermeture, το Ταμείο Αυτοεγγύσεως, καλύπτει εργαζόμενους που είναι σε τακτική βάση εργαζόμενοι στο Βέλγιο και επομένως αυτό καλύπτει απόλυτα αυτό το οποίο ζητάει η οδηγία παρά το γεγονός ότι ορισμένε φορές υπάρχουν δυσκολίε οι οποίε προκύπτουν, Παραδείγματο χάρη, όταν υπάρξει αφαιρεγγιότητα μια επιχείρηση σε ένα άλλο κράτο μέλος που επηρεάζει τους εργαζόμενους στο Βέλιο. Τότε είναι δύσκολο για το ταμείο αυτό, το de Fermeture, να πάρει τις απαραίτητες πληροφορίες από τους ε, υπευθύνους τι εταιρείας αυτής που είναι στο εξωτερικό για να ξέρει τι ακριβώς έχει γίνει ώστε να διακριβώσει αν πράγματι πρόκειται για περίπτωση πτώχευσης. Και αυτό είναι προβληματικό γιατί δεν υπάρχει εναρμόνιση των πτωχευτικών νομοθεσιών σε διάφορες χώρες και αυτό δημιουργεί προβλήματα για να πάρει τις σωστές πληροφορίες το Fond de αυτός αυτό το ταμείο αφήνει και περιθώριο ερμηνείας για τα κράτη-μέλη αυτή η οδηγία για το πώς θα πρέπει να καθορίζεται ο αρμόδιος φορέας για την παροχή εγγύησεων και από αυτή την άποψη ορισμένε φορές υπάρχουν πρακτικά προβλήματα. για τον καθορισμό των υπευθύνων. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η Πρόεδρος θα ήθελα να σας ζητήσω αν μπορείτε να μας αφήσετε τις παρεμβάσεις σας σε έγγραφη μορφή στην γραμματεία για να τις ε, διανύμουμε και στα μέλη της ε, Επιτροπής μας και τώρα ζητώ από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Φέντρας, αν μπορεί και θέλει να λάβει το λόγο από μέρους της Επιτροπής. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Η έκθεση που εξετάζεται σήμερα απορρέει από μια εξωτερική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ερωτηματολόγιο που έστειλε στις χώρες μέλη και στους κοινωνικούς εταίρους. Τους δόθηκε ευκαιρία επίσης και να σχολιάσουν τα αποτελέσματα της μελέτης. Η εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη-μέλη είναι το κύριο στοιχείο αλλά περιλαμβάνονται και άλλα στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό των εργαζόμενων που επωφελήθηκαν από τους οργανισμούς εγγύσεων κατά το παρελθόν. Για παράδειγμα, την περίοδο 2006 με 2009, 3,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι επωφελήθηκαν από τις πληρωμές αυτές, που δεν είναι και λίγο. Η έκθεση καταλήγει στο ότι οι διατάξεις έχουν εφαρμοστεί ορθά αλλά το ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες ανησυχίες όσον αφορά εφαρμοστικά μέτρα στα κράτη-μέλη. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να ελέγχει τη λειτουργία της οδηγίας αυτής από κοντά και θα χρησιμοποιεί ό,τι μέσα έχει στη διάθεσή της εφόσον εντοπιστούν προβλήματα. Ένα από τα άλλα συμπεράσματα της μελέτης τώρα. Αν δείτε την... το ιστορικό της οδηγίας αυτής, που είναι μεγάλο, δείχνει ότι εδώ και πάνω από 13 χρόνια πιστεύουμε ότι η οδηγία αυτή παίζει ένα ρόλο κλειδί, γιατί προσφέρει ένα ελάχιστο βαθμό προστασίας των εργαζόμενων μέσα στην εσωτερική αγορά. Ελάχιστος βαθμός προστασίας λοιπόν, πολύ σημαντικό. Και χάρη στην οδηγία αυτή, οι χώρες μέλη που δεν έχουν οργανισμούς εγγύσεων αναγκάστηκαν να τους δημιουργήσουν και τώρα παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις αφαιρεγκαιότητας και καλύπτουν τις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Συγχρόνως η μεταρρύθμιση ε, που έγινε μετά το 2002 αποσαφηνίζει τις νομικές διατάξεις στις διάφορες περιπτώσεις και προσαρμόζει τις προδιαγραφές ώστε να γίνονται αλλαγέ και στους νόμους περιφερειότητας των χωρών μελών και έτσι προσφέρει μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα στον κόσμο. Όσον αφορά τώρα τις διεκδικήσεις των κοινωνικών εταίρων. Ένα μικρό σχόλιο παρακαλώ. Τονίζω για άλλη μια φορά ποια είναι η φύση αυτής της οδηγίας. Η οδηγία αυτή προσφέρει έναν ελάχιστο βαθμό προστασίας. Αν κοιτάξετε για παράδειγμα το επίπεδο αμοιβών για το οποίο δεν μπορεί, δεν έχει την αρμοδιότητα η Επιτροπή να ρυθμίσει τίποτα, διαπιστώνεται ότι οι διαφορέ είναι μεγάλε μεταξύ των χωρών μελών. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά την περίοδο ευθύνη και το ύψο τη ευθύνη. Πάντως καθορίζοντα ένα ελάχιστο, αναρωτιόμαστε είναι αυτό ο καλύτερο τρόπο, γιατί ίσω έτσι τελικά καταλήξουμε σε μια ελάχιστη προστασία, η οποία είναι πραγματικά η χαμηλότερη δυνατόν και δεν είναι αυτή η θέση που θα θέλαμε εμείς να υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Ρέντου. Νομίζω ότι και με τη δική σας απάντηση μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν προβλέπει η Κομισιόν για το άμεσο μέλλον να παρουσιάσει μια τροποποίηση της οδηγίας αυτής. Νομίζω ότι από ό,τι κατάλαβα θα διατηρήσετε αυτή την πρόταση οδηγίας και θα έχουμε απλώ να αντιμετωπίσουμε το θέμα της εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε από το σημείο αυτού. Ίσως για να υπάρξει διευκρίνηση για το σημείο αυτό που ανέφεραν τα εκπρόσωποι των εργαζομένων, δεν υπάρχει καμιά πρόθεση να τροποποιηθεί η νομοθεσία, αλλά συγχρόνως η οδηγία αυτή αποτελεί τμήμα του λεγόμενου τεστ υγείας, όπως λέμε στην εσωτερική μας αργό. Αλλά για τα θέματα που αναφέρθηκαν έχουν να κάνουν οι οδηγίες της ε, και τη διαβούλευση με του εργαζόμενου. Αυτό είναι ένα τελείω διαφορετικό θέμα όμως. Εμείς έχουμε ξεκινήσει μόλις την ανάλυση αυτών των θεμάτων και ίσως το φως της κρίσης μπορεί να διαφανεί ότι σε ορισμένες πτυχές μπορεί να χρειαστεί να τροποποιηθεί αυτή η οδηγία ή θα μπορούσε να βελτιωθεί για να λειτουργεί καλύτερα. Αλλά όλη η άσκηση του τεστ υγείας και ευρωστίας συνεχίζεται ακόμα και αυτά που σας αναφέρω εδώ είναι μονάχα ένα μικρό τμήμα. Δεν θα έχουμε αποτελέσματα όμως μέχρι το τέλος του 2011 και θα υπάρξουν άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες μπορεί να είναι νομοθετικές αλλά όχι κατά ανάγκη νομοθετικές. Δεν προβλέπεται πριν από το 2013 δεν θέλουμε λοιπόν να τροποποιήσουμε αυτήν την οδηγία με το να θέσουμε ελάχιστα κατόφλια ή να νομοθετήσουμε σε σχέση με την έννοια των αποδοχών. Ποια πρέπει να είναι η συνολική έννοια των αποδοχών. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Νομίζω ότι ήταν σαφές αυτό το οποίο ήθελε να πει η Κομισιόν. Και τώρα μπορούμε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να λάβει το λόγο. Η κυρία Ρέγνερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ότι πρέπει λόγω της εσωτερικής αγοράς να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας των εργαζομένων. Και φυσικά αυτό πρέπει να περιλαμβάνει και περιπτώσει αφαιρεγκαιότητα των επιχειρήσεων στι οποίε εργάζονται. Υπάρχει και το θέμα των ε, ορισμών. Ξέρουμε ότι οι ορισμοί καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο και δεν είναι πάντα εναρμονισμένοι. Η οδηγία καλύπτει όλους αυτούς οι οποίοι εργάζονται στα κράτη-μέλη Και είπατε εσείς ότι στην εφαρμογή αυτής της οδηγίας υπήρξαν κάποια προβλήματα. Ιδίως με τον τρόπο μεταγραφής από τα κράτη-μέλη. Είπατε λοιπόν ότι υπάρχουν προβλήματα με την εφαρμογή των, ε, των συμβολέων εργασίας και δεν μπορούν να έχουν πλήρως τα την εφαρμογή των δικαιωμάτων του. Θα ήθελα να ξέρω στην περίπτωση της Τσεχίας πώς αξιολογείται αυτήν την ε, εξαίρεση η οποία δίδεται και αν δούμε καλύτερα την έννοια του εργαζομένου προφανώς περιλαμβάνει και μορφές ε, εργασίας ε, καθορισμένου χρόνου που καλύπτονται από την οδηγία αλλά το ερώτημα είναι αν αυτοί οι οποίοι είναι ασκούμενοι παραδείγματο χάρη, που είναι όλο και πιο δύσκολο ο καθορισμό αυτή τη έννοια του τι είναι κάποιο ασκούμενο, αν περιλαμβάνονται μέσα στην έκθεση αυτή και θα ήθελα να ξέρω πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα των ασκουμένων, που εδώ υπάρχει και μία πληθώρα εθνικών ορισμών. Επίσης, ένα άλλο ερώτημα αφορά ορισμένες μορφές εργαζομένων που είναι εκτός αυτής της ε, ε, οδηγίας, χάρη για τους ε, ναυτικούς ή για άλλες μορφές εργαζομένων. Υπάρχουν ίσως ιστορικοί λόγοι για κάτι τέτοιο, αλλά αναρωτιέμαι αν είναι πράγματι σωστό να βρούμε έναν τρόπο να τους συμπεριλάβουμε όλους αυτούς τους εργαζομένους. Και μια τρίτη ερώτηση την οποία θα ήθελα να θέσω εγώ αφορά την περίπτωση, την περίπτωση πτωχεύσεων που καλύπτουν διαμεθοριακά εργαζόμενους και αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται όλο και περισσότερο στην Ευρώπη. Όλο και περισσότερο αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό των διαμεθοριακών σχέσεων. Είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο πια. Προβλέπει η οδηγία μια ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και θέλω να θέσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα τώρα προς την Κομισιόν. Μήπως θα ήταν πιο χρήσιμο να υπάρξει μια τροποποίηση που θα οδηγήσει στο να είναι υποχρεωτική η παροχή πληροφοριών σε περίπτωση διαμεθοριακής εργασίας να εξασφαλιστεί λοιπόν αυτό ότι θα μπορούν να υπάρχουν οι πληροφορίες σε διαμεθοριακό επίπεδο για επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα τα οποία είναι διαμεθοριακοί εργαζόμενοι. Ευχαριστώ αυτά. <coughs> Ευχαριστώ πολύ. Άλλοι δύο μιλητέ. Η κυρία Στάινμπρουκ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο ορισμός του τι είναι αποδοχές νομίζω ότι εμπίπτει στο εθνικό δίκαιο της κάθε χώρας. Και αυτό είναι Κάτι το οποίο οδηγεί σε διαφορετικές ε, παροχές από τα ταμεία εγγύσεων. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί τώρα αυτό το θέμα <clears throat> προς την Κομισιόν το ερώτημα. Και τέλος, ο κύριος Μπόλοντ έχει το λόγο. Ναι, για το ΕΛΚ ε, με μια έκθεση βάση της διαβούλευσης με την Επιτροπή και της έκθεσης του κ. Ζέρλινγκ ε, εργάστηκα και η οδηγία 2008 που νομίζω ότι είχε αποδείξει ότι είναι υπέρ αυτής της ε, προστασίας σε περίπτωση αφεργιώτας. Όπως είπαν και διάφοροι εδώ μιλητές οι προηγούμενοι, όσοι έλαβαν τον λόγο, βλέπουμε τα κενά αυτές τις οδηγίες, ε, κάποια κενά και αντιμετωπίζουμε προβλήματα ορισμού βέβαια και επικουρικότητας. Πολλά κενά εναρμόνιση υπάρχουν στα κράτη-μέλη πάνω σε όρους ε, που δεν μπορούν να παρακαμφθούν και για να επιτρέψουν μια εναρμόνιση και για να υπερασπιστούμε όσο γίνεται καλύτερα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτά είναι ο ορισμός του εργαζόμενου, του μισθωτού, της αμοιβή του μισθού, όπως είπαμε, την περίοδο αναφοράς ποια είναι αυτή και επίσης υπάρχει ένας ορισμός από πότε ισχύει αυτή η αφαιρεγγιότητα, πότε όταν κάποιος κηρύσει πτώχευση, μάλλον ζητάει την πτώχευση είτε την πραγματική περίοδο τι γίνεται, προσπαθήσαμε να δούμε ανάλογα με διάφορε προτάσει. Η Επιτροπή λέει ότι δεν θα ήθελε στο σημείο αυτό να αλλάξει την οδηγία και παρα, παραμένοντα από τη στιγμή που πρόκειται για ένα πλαίσιο οικονομική κρίση, ακόμα μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα και γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να προσθεθεί προτείνουμε ρυθμίσεις, ε, γι' αυτό ακριβώς προτείνουμε περίπου 20 τροπολογίες βάσει της ε, έκθεσης κυρία Ζέρλιν για μια καλύτερη εναρμόνιση και υποβάλλοντας προτάσεις για μια ελάχιστη αποζημίωση για τους μισθωτούς και επίσης ένα περιθώριο, μάλλον το όριο παρέμβασης, ε, τι γίνεται ακριβώς όσον αφορά την αφαιρεγγιότητα και μέσω αυτών των τροπολογιών παρεμβαίνουμε, υποβάλλουμε προτάσεις και έτσι όσοι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν παρόμοιες περιπτώσεις ή θα αντιμετωπίσουν ε, ενδεχόμενα να, μπορέσουμε να μπορέσει κανείς να τους περασπιστεί όσο γίνεται καλύτερα και να μην μπερδέψουν με διοικητικά εμπόδια που θα προσθέσουν ακόμα περισσότερα προβλήματα στα δικά του ε, ήδη υπάρχοντα επαγγελματικά προβλήματα. Αυτό δεν θα επιστρέψει σε λεπτομέρειε όσον αφορά τις προτινόμενε τροπολογίε, αλλά πρόκειται για δρόμους προσανατολισμού για να βελτιώσουμε το πλαίσιο τη σημερινή οδηγία. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι δεν θέλει κανείς άλλος να ζητήσει το λόγο. Τότε θα δώσω το λόγο στην στους εκπροσώπους και πάλι των ε, <clears throat> κοινωνικών εταίρων της Ευρωπαϊκής ε, Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, αν θέλουν να προσθέσουν κάτι, και πάλι στην Κομισιόν μετά, στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Θέλετε να πείτε κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας όσον αφορά τον ορισμό. Τι είναι εργαζόμενος και ποια κατάσταση επικρατεί στην Τσεχία. Ακόμα και η οδηγία όσο έχει τώρα. Οι ορισμοί δηλαδή που έχουμε ήδη στην οδηγία επιτρέπουν στην Τσεχία να το συμπεριλάβει στην προστασία από την οδηγία αυτή. Οπότε μπορεί να υπάρξει παραβίαση της οδηγίας και δηλαδή θα ήταν δυνατόν να αναλυφθεί η δράση ήδη και σήμερα κατά της Τσεχίας. Ακόμα και αν δεν υπάρξει αλλαγή. Αλλά υπάρχει πάντα το γενικό ζήτημα του πώς ορίζεται ο εργαζόμενος, τι είναι εργαζόμενος. Αναφερθήκατε σε διάφορα προβλήματα. Αναφερθήκατε στο πρακτικό ζήτημα, σε ορισμένε χώρε καλύπτονται, σε ορισμένε για τους μαθητευόμενους, τους ασκούμενους. Υπάρχει το πρόβλημα των οικιακών βοηθών. Ξέρουμε ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στην Ευρώπη. Πάντα δηλαδή πέφτουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα του τι σημαίνει εργαζόμενος για την κάθε χώρα μέλους. Είναι ένα γενικό πρόβλημα, όπως σας είπα, και δεν πρόκειται να λυθεί με την οδηγία για την Αυθαιρεγκαιότητα. ίσως ένα βαθμό να λυθεί ε, μέσω κάποιας άλλης νομοθετικής πράξης. Μια άλλη ερώτηση ήταν οι διαφορές στις πληρωμές. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιες διαφορές. Για μας το πιο σημαντικό είναι να πούμε ότι αν υπάρχουν διεκδικήσεις των εργαζόμενων, πρέπει να καλυφθούν. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση ε, μέσω μιας ευρωπαϊκής οδηγίας. Όχι. Όπως είπα και πριν, για μας ο πραγματικός στόχος είναι πώς θα οριστεί ο εργαζόμενος στην οδηγία και πώς θα ενσωματωθεί αυτό στην εθνική νομοθεσία. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Να συμπληρώσω κι εγώ, λέει ο κύριος Φαντεμπέρκ, για τις διασυνοριακές περιπτώσεις. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι ούτε και εδώ έχουμε κάποια ξεκάθαρη απάντηση, γιατί το θέμα έχει να κάνει με το εμπόριο και δεν μας αρέσει και πολύ να παρεμβαίνουμε. Όμως υπάρχει το πρόβλημα ότι οι διαδικασίες φερεγγιότητας είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα και σε περίπτωση φερεγγιότητας μιας διασυνοριακής επιχείρησης οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στα διάφορα κράτη, διαφορετικές μεταξύ τους όπως είπαμε, ενδιαφέρουν μεταξύ τους. Γιατί ακολουθούν την νομοθεσία στην κάθε χώρα. Οπότε οι οργανισμοί εγγύησης ε, δυσκολεύονται να έχουν πληροφορίες. Πρέπει να έχουν πληροφορίες από τα δικαστήρια των διαφόρων χωρών. Άρα πρέπει να δούμε πώς οι πληροφορίες αυτές μπορούν να προχωράνε πιο γρήγορα, να ανταλλάσσουν αυτές τις πληροφορίες οι χώρες μέλη μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Κομισιόν. Έχετε τρόπο κύριε Φέντρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Τα, τα παραδείγματα που δώσατε είναι ακριβώ αυτά που βρίσκεται στι σελίδε 1 και 2. Αναφέρεται η περίπτωση τη Τσεχία, αναφέρεται η Κύπρος Αυτά είναι κυρίως τα προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί και προσπαθούμε να λύσουμε σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Για το διασυνοριακό ζήτημα, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο εξής. Ένα από τα κύρια στοιχεία της πρότασης του 2002 που συμπεριλάμβανε την ε, υπερεθνική περίπτωση μιλούσε για συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών. Πηγαίνετε στη σελίδα 6 της έκθεσης. Θα δείτε εκεί ότι έχουμε ένα εντυπώ στάνταρτ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανταλλαγή πληροφοριών. Άρθρο 11, αλλά και ανταλλαγή πληροφοριών για τις ανώτατες ποσότητες που προβλέπονται στην Εθνική Νομοθεσία. Αυτά είναι τα άρθρα 4.1 και 4.3. Αυτά, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Γκέρλινγκ, αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στα αγγλικά λέμε αν κάτι δεν έχει σπάσει να μην πάμε να το ξανακολλήσουμε. Ό,τι λειτουργεί πρέπει να το αφήσουμε όπως έχει. Χαίρομαι που υπάρχει μια γενική συμφωνία εδώ για την οδηγία και είναι χρήσιμο να ξέρουμε ότι στο Βέλιο τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος, το 90% των διεκδικήσεων ικανοποιούνται. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτό το λόγο τους κοινωνικούς εταίρους για την παρουσία τους και για το γεγονός ότι σε μεγάλο βαθμό επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία έχω ε, ανακαλύψει στις δικές μου άτυπες επαφές πριν συντάξω <clears throat> αυτήν τη γνωμοδότηση. Ξέρω ότι παραμένουν κάποια θέματα τα οποία δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε, αλλά τα θέματα αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με τη μεταγραφή της οδηγίας και την εφαρμογή της. Χαιρετίζω ιδιαίτερα την δήλωση της Κομισιόν σχετικά ότι κοιτάνε προς κοιτάνε τα θέματα αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα της γνωμοδότησής μας να περιλάβει, να διαλάβει τα θέματα αυτά. Απλώς έχω ένα βασικό πρόβλημα με την ιδέα του να προταθεί ένα ελάχιστο επίπεδο αποζημίωσης, όχι μόνο γιατί αυτό θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο στην πράξη με 27 κράτη-μέλη, θα μπορούσα να φανταστώ <clears throat> ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια μαθηματική, ένας μαθηματικός τύπος και όχι ένα συγκεκριμένο ποσό που να καλύπτει όλους, ακόμα και αυτό θα ήταν δύσκολο κάτω από τις τωρινές συνθήκες. Πιστεύω ότι το σύνολο θέμα του χαμηλότερου κοινωνικού, του χαμηλότερου κοινού παρονομαστή είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για πολλά κράτη-μέλη, γιατί πολλά κράτη-μέλη δίνουν πολύ περισσότερη αποζημίωση από ό,τι φαντάζομαι θα καταλήγαμε σε περίπτωση μιας κοινή αποζημίωσης και είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα το να θέλουμε να έχουμε ένα κοινό μεσονόρο, γιατί αυτά τα κράτη-μέλη που πληρώνουν περισσότερο θα υποχρεωθούν να κατέβουν προς τα κάτω. Τέλος, να αναφέρω και πάλι τα θέματα τα διαμεθοριακά. Νομίζω το είπαμε προηγουμένως στην ανταλλαγή απόψεων που είχαμε πριν από ένα μήνα, ότι ο στόχος μου είναι να καταθέσω και τις δικές μου τροπολογίες στη γνωμοδότηση αυτή, διότι αποκόμισα και περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα αυτά και πιστεύω ότι χρειάζεται, έχοντας δει την έκθεση της Κομισιόν, να καλύψουμε ένα ουσιαστικό θέμα για τους ε, εργαζόμενους όταν πρόκειται για την ε, θέση σε προτεραιότητα των πιστωτών. Πρέπει να έχουν ένα, να υπάρχει μια κοινή ιεραρχία για την ικανοποίηση των πιστωτών μιας εταιρείας που έχει πτωχεύσει. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει και η νομική υπηρεσία να έχουμε μια σαφή θέση των εργαζομένων στην ιεραρχία διεκδικήσεων έναντι μιας εταιρεία η οποία έχει πτωχεύσει. Θα πρέπει λοιπόν να το κάνουμε αυτό για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε μερικά από τα προβλήματα που προκύπτουν για την προστασία των διαμεθοριακών εργαζομένων. Σας ευχαριστώ λοιπόν και κλείνω σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους αυτούς που έλαβαν το λόγο και ιδίω του καλεσμένου μα από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων και την Κομισιόν. Και θέλω απλώ να κάνω το εξή σχόλιο για αυτά που είπε η κυρία Γκέρλινγκ, την τελευταία δήλωση της κυρίας Γκέρλινγκ, για την πρόταση αυτή, για την ιεράρχηση των πιστωτών των επιχειρήσεων. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Στην ίδια μου τη χώρα, στην Πορτογαλία, προκύπτουν πολλές φορές προβλήματα με αυτό το θέμα. και αν σε ορισμένε περιπτώσεις τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί υπέρ των εργαζομένων, δίνοντάς τους προτεραιότητα στην καταβολή των, ε, των οφειλωμένων σε περίπτωση αφαιρεγγιότητος μιας εταιρείας, σε άλλες περιπτώσεις δεν έγινε αυτό. Και δόθηκε η προτεραιότητα στο κράτος ή στις τράπεζες. Και οι εργαζόμενοι έμειναν στον Άσο. Γι' αυτό το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιτύχουμε η οδηγία αυτή να δώσει μια σαφή απάντηση στο θέμα αυτό και φυσικά <clears throat> είναι και, πρέπει να είναι και σημείο μέρημνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω δει σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι να θίγονται λόγω αυτής της ε- έλλειψης μιας ιεραρχίας σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση των ε, διεκδικήσεων για μια αφαιρέγγια εταιρεία. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να τονίσω ότι συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη της κυρίας Γκέρλινγκ. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Θα περιμένουμε λοιπόν την επόμενη φάση των προτάσεων τροπολογίας. Και έχουμε κλείσει και αυτό το σημείο τώρα. então, eh, Επομένως, μετά από τις ε, αλλαγές που έχουμε κάνει στην ημερήσια διάταξη, θα περάσουμε τώρα στο σημείο 5, δημογραφική αλλαγή και οι συνέπειέ τη για την μελλοντική πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εισηγήτρια είναι η κυρία Σαρία Σταγιά, που είναι παρούσα πλέον και βεβαίως θα μας ομιλήσει για τις απόψεις της σε σχέση με τις τροπολογίες και τις προτάσεις συμβιβαστικού χαρακτήρα για τις, την ψηφοφορία που θα γίνει αύριο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Έχω πει και άλλη φορά ότι εδώ στην Επιτροπή μας είχαμε μια πολύ πλήρη έκθεση για τις δημογραφικές αλλαγές. Στη γνωμοδότησή μας λοιπόν εδώ χειριζόμαστε τις αλλαγές που έχουν γίνει και πώς επηρεάζουν την πολιτική συνοχή. Δηλαδή περιοριζόμαστε μόνο σε αυτό το θέμα της δημογραφικής αλλαγής και της νέπιές τη στη μελλοντική πολιτική συνοχή. Ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής αυτής που υπέβαλαν τροπολογίες. Πολλές τροπολογίες μάλιστα. Είναι όμως πολύ επικοδομητικές Βοηθάνε πολύ την έκθεση, τη βελτιώνουν. Έχουμε καταλήξει σε τέσσερις συμβιβαστικές προτάσεις. Και θα υπάρξουν και τέσσερις κατατμήματα ψηφοφορίες. Μία ζήτησε το ΕΛΚ, δύο η ΓΚΟΕ και μία κατατμήματα ψηφοφορία ζήτησαν οι πράσινοι. Θέλω να σχολιάσω λίγο Πρώτα απ' όλα την τροπολογία 43 και την κατατμήματα ψηφοφορία που ζήτησε η δικιά μου ομάδα, το ΕΛΚ. Έχει να κάνει με μια πρόταση που λέει ότι ζητάει από την Επιτροπή να διασφαλίσει την νομική βεβαιότητα των υπηρεσιών ε, κοινοφελών υπηρεσιών, των επιχειρήσεων κοινοφελών υπηρεσιών και να τηρηθεί επικουρικότητα. Γι' αυτό ζητάμε κατατμήματα ψηφοφορία εδώ. Έπειτα υπάρχει και η τροπολογία 31 της κυρίας Φλέτσε. Στην τροπολογία αυτή θέλει να αντικατασταθεί όρος παραγωγικότητα από τον όρο προσβασιμότητα. Ποιο είναι το νόημα. Το νόημα αλλάζει ουσιαστικά και γι' αυτό ακριβώς και είμαι κατά της αλλαγής αυτής. Εγώ θα ήθελα να είμαστε, να βοηθάμε και όχι να δημιουργούμε περισσότερες δυσκολίες. Τέλος πάντων είναι σημαντικά και τα δύο αυτά θέματα, αλλά εγώ όπως σας είπα έχω βάλει πλην εκεί δίπλα στην τροπολογία αυτή. Τώρα οι πολιτικές ομάδες που ζήτησαν τις άλλες κατά τμήματα ψηφοφορείς ίσως θα μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί και να πούνε ποια είναι η δικιά τους θέση από αυτόν. Γιατί ζητάνε καταδημάτα ψηφοφορία. Αλλιώς, το μόνο που έχω να πω είναι ότι είναι πολύ πικοδομητική η γνωμοδότηση αυτή και πιστεύω ότι η Επιτροπή μας θα βοηθήσει να προχωρήσει καλά η έκθεση που έχει αναλάβει η Ρέγγι. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ λέει και η κυρία Φιγκεϊρέντο, κυρία Βουλευτής. Και τώρα είναι ανοιχτό το πεδίο για συζήτηση. Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος θα ήθελε να κάνει κάποια παρατήρηση ή να θέσει κάποιο ερώτημα. Κυρία Οβίρ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Σάρη Εσάια για την σαφή διατύπωση που έχει το εγγραφό της, για τη σαφήνεια της γνωμοδότησής της. Και νομίζω ότι λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη στην γνωμοδότησή τη. Η πολιτική μου ομάδα των φιλελευθέρων είναι πολύ ικανοποιημένη με αυτή την ε, γνωμοδότηση και γι' αυτό έχουμε καταθέσει μόνο τρεις τροπολογίες. Τις υποστηρίζει η Σιγίτσα και γι' αυτό θέλω να την ευχαριστήσω και θέλω να ευχαριστήσω όλου αυτούς οι οποίοι έχουν συμβάλει στην σύνταξη αυτού του εγγραφού. Ευχαριστώ. η κυρία Σρόντερ. Συγγνώμη. Αλλά ήμουνα σε μια διαβούλευση για την πέμπτη ε, έκθεση συνοχής. Θα ήθελα μονάχα να αναφερθώ σε ένα σημείο. Θα θέλαμε να υπάρχει μια προφορική τροπολογία που θα καταθέσουμε για την τροπολογία 19, μια προφορική τροποποίηση λοιπόν που αποσαφηνίζει ότι ο στόχος είναι να γίνουν πιο ενεργοί οι ηλικιωμένοι ώστε να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας γιατί η, Φιλανδία, η αγγλική ε, διατύπωση εμπνέεται από το φιλανδικό σύστημα το οποίο είναι πολύ καλό για τη Φιλανδία που έχει μια παράδοση για τα θέματα αυτά αλλά δεν είναι ίσως η καλύτερη διατύπωση για άλλα και δεν είναι ίσως η καλύτερη διατύπωση για να καλύψει όλους. E Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θέλει να λάβει το λόγο. Και δίνω και πάλι το λόγο στην κυρία Εσαΐα, εάν θέλει και πάλι να πει κάτι. Για να κλείσουμε και αυτό το σημείο. Ελπίζω ότι αύριο δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα με την ψηφοφορία, αλλά αν υπάρξει αυτή η προφορική τροποποίηση πρόταση τροπολογίας θα ήταν χρήσιμο να την έχω προηγουμένως γραπτός, ώστε να δούμε αν ε, είναι μεταφραστικού χαρακτήρα, είναι γλωσσικού χαρακτήρα αυτή η τροπολογία ή αν είναι θέμα ουσίας. Στην Φινλανδία έχουμε πολύ θετικά κίνητρα για τους ανθρώπους που θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται και να έχουν μια μακρύτερη χρονικά καριέρα. Και αυτά τα κίνητρα λοιπόν λειτουργούν ώστε αυτοί οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν στην ε, εργασία μπορούν να το κάνουν και αποκομίζουν και κάποιο κέρδος και αυτό είναι ένα διαφορετικό σύστημα από άλλες χώρες όπου μαστιγώνονται αυτοί οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται. Στη Φιλανδία αντίθετα τους παρέχουμε κίνητρα. Αλλά αν έχετε έτοιμη αυτή την προφορική τροπολογία είμαι έτοιμη να τη συζητήσω μαζί σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ λαϊκή Πρόοδο. Έχει κλείσει λοιπόν και το ζήτημα αυτό. Και το επόμενο είναι το σημείο 8, η πρόθεση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι εδώ είναι παρόν ο κύριος Ουγγουριάνου. Και δεν ξέρω αν θα θέλατε να λάβετε το λόγο για το ζήτημα αυτό, για την εκθεσή σας, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να συζητήσουμε για τις ε, νομοδοτήσεις που έχουν κατατεθεί από διάφορους συναδέλφους. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 157 τροπολογίες που δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον από τα μέλη της Επιτροπής μας. Είμαι πολύ ικανοποιημένο που παίρνει μορφή η έκθεση σιγά σιγά. Είναι σαφές ότι όλοι συμφωνούν, οι περισσότεροι συμφωνούν, ότι χρειαζόμαστε αυτή την κινητικότητα των εργαζομένων και χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερη κινητικότητα εργαζομένων. Υπάρχει όμως ένα διαδικαστικό ζήτημα από την αρχή, ε, μικρή σημασία ίσως, είναι ότι πρέπει να υπάρχει μία ενότητα για αυτή την ε, έκθεση από πλευράς τεχνολογίας, από πλευράς ε, όρων. Πρέπει να χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις για να λέμε το ίδιο πράγμα. Ο, είτε πρόκειται για τους μετανάστες, ε, αν εννοούμε Ευρωπαίους, αν εννοούμε άλλους. Πρέπει να ξέρουμε τι εννοούμε με τους όρους που χρησιμοποιούμε και να εννοούμε όλοι το ίδιο. Κατόπιν τούτον με ικανοποιούν πολύ οι ιδέες των τροπολογιών. Μιλάνε για ίδιους μισθούς για ίδια απασχόληση, ανεξάρτητα με το πού είναι αυτή η απασχόληση. Δεύτερον, θέλουν να αποφεύγουμε το κοινωνικό dumping. Τρίτον, μιλάνε για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας. μιλάμε για εργαζόμενους και το δικαίωμα στην εργασία. Τέταρτον, διασφάλιση θέσεων απασχόλησης και συνθήκων εργασίας. Για να μιλήσουμε τώρα πιο συγκεκριμένα για τις τροπολογίες. Θέλω να αναφερθώ στις τροπολογίες που προωθούν την ιδέα της αναγνώρισης των διπλωμάτων και των προσόντων για τους πολίτες είναι ζωτική σημασία σε αυτό. Οι συνάδελφοι Χάρκιν και Σαρτιέ, Χαρτιέ, Κάμπερνοφ έχουν υποβάλει τροπολογίες γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα της αναγνώρισης. Μία άλλη πτυχή έχει να κάνει με τροπολογίες όσον αφορά το Solvit και το Eures, που είναι ζωτική σημασίας μέσα εργαλεία. Αν θέλουμε κινητικότητα των εργαζομένων και να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε ε, χαίρομαι πολύ για τις τροπολογίες αυτές που μιλούν για τη σημασία που έχουν οι Solvit και οι Eures. Κάτι άλλο ενδιαφέρον είναι η ιδέα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες να χρησιμοποιούν και να χαίρουν πλήρως των δικαιωμάτων τους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει πολύ. Και για την εθνική νομοθεσία και για την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μιλάω εδώ για την τροπολογία αριθμός 15 του κύριου Κάμπερνοχ. Υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες που τονίζουν τη σχέση των πολιτικών για την εργασία και άλλων πολιτικών, για την υγεία των εργαζομένων, για παράδειγμα, η αποφυγή διπλής φορολόγησης ή άλλα προβλήματα που μπορούν να αποτρέψουν τους εργαζόμενους στην κινητικότητά τους. Όταν μιλάμε για κινητικότητα των εργαζομένων πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η κινητικότητα αυτή μπορεί να δημιουργήσει κάποιες αρνητικές καταστάσεις. Αρνητικές τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες. Κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα πρέπει να αναφέρονται και τέτοια πράγματα πρέπει να αναφέρονται εδώ και τα αναφέρει ο Σκιώδης εισηγητής από τους σοσιαλιστές. Ένα άλλο θέμα τώρα έχει να κάνει για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την κινητικότητα των εργαζομένων. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι σωστή η ευρωπαϊκή προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορώ να δεχτώ τροπολογίες που προωθούν την ιδέα που λέει ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση δεν είναι σωστή. Τροπολογίες που λένε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν έχει φτιαχτεί για να υποστηρίξει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν είναι σωστή. Δεν μπορούμε να επιχειρηματολογήσουμε για κάτι τέτοιο. Ένα άλλο ενδιαφέρον πρόβλημα εδώ, που το είδα σε διάφορες τροπολογίες, είναι η ιδέα της μετανάστευσης των εργαζομένων όταν δεν γίνεται στη θελοντική βάση. Δηλαδή υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες υπονοούν ότι αναγκάζονται εργαζόμενοι να μετακινηθούν, να ψάξουν δουλειά αλλού. Χωρίς να αρνούμαστε την, την οικονομική πίεση ή το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε, η Ευρώπη γενικά και κυρίως η Νότια Ευρώπη, παρόλα αυτά θα έλεγα ότι η κινητικότητα αυτή γίνεται σε θελοντική βάση και όχι καταναγκαστικά. Υπάρχουν και μερικές τροπολογίες που αναφέρονται σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι μετανάστες Τούρνεν, Κορνέλισεν έχουν τέτοιες τροπολογίες όπου τονίζουν ότι πρέπει να δούμε το θέμα της ε, παράνομης εργασίας και τι δράσεις μπορούν τι δράσεις μπορούν να ληφθούν για να χαίρουν οι μετανάστες πλήρως των δικαιωμάτων τους στις χώρες που πηγαίνουν. Τέλος, την έκθεση αυτή εγώ την βλέπω όχι σαν μία βραχυπρόθεσμη συνταγή, μεσοπρόθεσμη, όχι, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να επηρεάσει και τις ε, χώρες που θα ενταχθούν μελλοντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κινητικότητα των εργαζόμενων, όπως είπα και νωρίτερα, μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες αρνητικές επιπτώσεις. Αλλά, αλλά, ξέρουμε ήδη από την πρόσφατη εμπειρία μας ότι τα θετικά είναι παραπάνω από τα αρνητικά. Και έτσι πρέπει να έρθουν όλοι οι φραγμοί. για να μπορούν οι εργαζόμενοι να βρουν δουλειά όπου ψάχνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χαίρομαι για την απόφαση που θα λάβει η Αυστρία και η Γερμανία, όπου η Γερμανία θα τους φραγμούς που είχε θέσει το 2004. Τέτοιου είδους φραγμοί όντως πρέπει να καταργηθούν και για τις χώρες που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και περιμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ λέει και η Πρόεδρος. Έχουμε ήδη κάποιους ομιλητές. Θα ήθελα όμως απλώς να προσθέσω ότι υπήρξαν δύο γνωμοδοτήσεις που ζητήθηκαν από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και υπάρχουν και 157 τον αριθμό τροπολογίες, 24 εκ των οποίων του ιδίου του εισηγητού. Βρισκόμαστε τώρα στα πλαίσια της συζήτησης. Η κυρία Βολινκιασέτε έχει ζητήσει το λόγο. Είναι εκεί. Πού είναι. Έχετε το λόγο και νομίζω ότι είσαστε ε, συντάκτρια γνωμοδότηση στην Επιτροπή Δημοσίου Ελευθεριών, Λίμπε. Έχετε το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ. Ακούστε. Είμαι η συντάκτρια γνωμοδότηση στην Επιτροπή ε, Δημοσίου Ελευθεριών και σκιώδης εισηγήτρια για την ομάδα των σοσιαλιστών και θα ήθελα να εκφράσω τη δική μου άποψη ευχαριστώντας πρώτα τον εισηγητή, τον κύριο Ουγγουρεάνου, για το έργο που έχει φέρει σε πέρας και για το σχέδιο έκθεσης. Νομίζω ότι ο εισηγητής έχει καταθέσει μια σειρά από προτάσεις και εάν μπορέσουμε να τις εφαρμόσουμε τις προτάσεις αυτές θα επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα και θα αρθούν τα εμπόδια για την διακίνηση, την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούν λοιπόν να ψάξουν για εργασία σε άλλες χώρες διατηρώντας πλήρως τα δικαιώματά τους. Θέλω επίσης να παρουσιάσω και ορισμένε εξηγήσει σε σχέση με τις τροπολογίες που έχουμε καταθέσει στην έκθεση του κυρίου Ουγγουριάνου. Πρώτα απ' όλα, για ένα γενικό σχόλιο η κινητικότητα του, των εργαζομένων, η ελεύθερα επιλεγόμενη κινητικότητα των εργαζομένων είναι ένα θετικό φαινόμενο και το έχει τονίσει ο εισηγητής. Στην τροπολογία μου όμως εγώ, στις τροπολογίες μου, θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τον αρνητικό αντίκτυπο της κινητικότητας των εργαζομένων. Δεν πρέπει να το παραγνωρίσουμε αυτό ούτε να το φοβόμαστε. Όχι μόνο να εξετάσουμε την τωρινή κατάσταση, αλλά να κοιτάξουμε και το μέλλον δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι στις χώρες της κεντροανατολικής Ευρώπης τα επίπεδα μετανάστευσης είναι πολύ υψηλά. Οι πολίτες μας μετακινούνται σε άλλα κράτη-μέλη. Μεταναστεύουν σε άλλες χώρες μέλη ελεύθερα, αλλά το πραγματικό κίνητρο πίσω από αυτή τη μετανάστευση είναι η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης στην ίδια την πατρίδα τους. Πρέπει να άρουμε λοιπόν όλα τα εμπόδια και όλους τους φραγμούς που υπάρχουν ήδη στις χώρες αυτές της κεντροανατολικής Ευρώπης. Υπάρχουν κάποια χωριά στις κεντροανατολικές ευρωπαϊκές χώρες όπου έχουν αδειάσει, έχουν φύγει όλοι οι άλλες περιοχές και άλλες χώρες. Και επομένως ο αντίκτυπος της ε, ε μετανάστευσης μπορεί να έχει και ένα αρνητικό χαρακτήρα. Ένα άλλο σημείο που θέλω να τονίσω, που είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών έχει να κάνει με τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει μια σειρά απονομοθετήματα, τα οποία στοχεύουν στο να εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των <clears throat> εργαζομένων, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. Να έχουν λοιπόν κοινά εργατικά, εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Δεν φτάνει όμως η νομοθεσία. Είναι το θέμα της εφαρμογής και της αστυνόμευσης της εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας. Θα πρέπει να μην σκεφτούμε μόνο τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά τα εφαρμοστικά μέτρα με τα οποία εξασφαλίζονται τα δικαιώματα αυτά και σε περιπτώσεις παραβιάσεων θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός επιφολής κυρώσεων και ε, θεραπείας των αδικαίων αυτών. Ο κύριος Ουγγουρεάνο έχει πει ότι συμφωνεί με τέτοιες τροπολογίες. Ένα άλλο κομμάτι των τροπολογιών μου αφορά την παρακολούθηση της, των επιθεωρήσεων εργασία στα κρατη Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία για να εξασφαλίζεται ότι οι εργασιακοί συμβάσεις είναι σύμμορφες με το όχι μόνο με το εθνικό αλλά και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία επίσης και σε σχέση με τα γραφεία ευρέσεως εργασίες και θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας στο να αυξήσουμε την συνειδητοποίηση για τα θέματα αυτά και να υπάρχει καλύτερη παροχή πληροφοριών προς τους εργαζομένους. Και θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε και τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων με τις εργατικές ενώσεις και συντεχνίες. Γιατί αν δεν υπάρξει αυτή η στενή συνεργασία, τότε τα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων θα φύγουν ή θα μπορούσαν να φύγουν. Και αυτό δεν προσθέτει στα θετικά στοιχεία της κινητικότητας της εργασίας. Μία ακόμα τροπολογία. Έχει να κάνει με την εφαρμογή της λεγόμενης οδηγίας περί πληροφορήσεως. Πολλές φορές οι μεταναστεύοντες εργαζόμενοι την χάνουν παραβιάσεως των δικαιωμάτων τους γιατί ο εργοδότης δεν τους πληροφορεί για το εργασιακό δίκαιο που ισχύει στη χώρα που εργάζονται και βρίσκονται οι εργαζόμενοι αυτοί σε αποδυναμωμένη θέση, γιατί δεν ξέρουν ίσως και τη γλώσσα του κράτους στο οποίο εργάζονται και πολύ πιθανό να μην γνωρίζουν και το εργασιακό δίκαιο. Αυτές λοιπόν οι τροπολογίες μου και ελπίζω θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε επιτυχώς και στο μέλλον με τον εισηγητή για την έγκριση αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λέει και η Πρόεδρος και δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Τούρνεν. Um, uh, Ευχαριστώ. Έρχομαι από την εσωτερική αγορά και υποθέσει καταναλωτών από αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Εκεί ο Επίτροπος Μπαρνιέ μόλις παρουσίασε τον κατάλογό του για την εσωτερική αγορά, γιατί έχει εκεί μια πρόταση, την αριθμός 10, για την κοινωνική συνοχή, την απόσπαση εργαζομάτων, και μιλάει εκεί και για τα κοινωνικά δικαιώματα, πώς να διασφαλίσετε δηλαδή η εφαρμογή των κοινωνικών δικαιωμάτων. Δηλαδή και σε εκείνη την Επιτροπή αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν προκλήσεις όταν συζητάμε για εργαζόμενους που δουλεύουν σε άλλη χώρα από τη δικιά τους και ότι υπάρχουν προκλήσεις, δυσκολίες όσον αφορά τους αποσπασμένους εργαζόμενους και πρέπει να κάνουμε διευκρινήσεις σχετικά με τα προβλήματα αυτά. Αυτό είναι ένα το οποίο ίσως θα έπρεπε να συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, αλλά έχει άμεση σχέση με αυτή την έκθεση. Ξεκινάω ευχαριστώντας τον εισηγητή. Θέλω να εξηγήσω λιγάκι τις τροπολογίες μας, γιατί ρωτήσατε κάποια πράγματα για τις τροπολογίες των πρασίνων. Έχουμε λοιπόν κάποιες τροπολογίες που μιλάνε για την αυταπασχόληση, μάλλον για την καταναγκαστική ε, μετανάστευση. Εδώ δεν εξετάζεται παρκώς με την έκθεση αυτή αυτό το θέμα. Ο κίνδυνος δηλαδή εκμετάλλευση των ανθρώπων αυτών. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα από τα συνδικάτα που μου διηγούνται ιστορίες, οι οποίες σοκάρουν για την ε, κακομεταχείριση των ανθρώπων αυτών. Είναι μια ομάδα κινδύνου που πρέπει να έχουμε υπόψη μας και να τους προστατεύσουμε. Έχουμε υποβάλει και μια τροπολογία, την 69, που μιλάει για την πρόσβαση στις κοινωνικές ε, παροχές. Και τι λέει. Λέει ότι αντί να περιοριστεί αυτή, αυτό το δικαίωμα στις κοινωνικές ε, παροχές, Ξέρω ότι εσείς θέλετε παραδείγματα. Το Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν μέχρι τώρα είχε ένα κανόνα που έλεγε ότι οι εργαζόμενοι που έρχονται από τις ανατολικές ε, χώρες δεν έχουν καθόλου δικαίωμα σε, κοινωνική, σε κοινωνικά δικαιώματα τον πρώτο χρόνο παραμονής του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέτοιες πολιτικές είναι που εμείς ε, καταδικάζουμε και 69 η τροπολογία μας λέει ότι ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται για τα δικαιώματα που έχει και για την πρόσβαση που μπορεί να έχει στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Η τροπολογία μας 103 επίσης μιλάει για την κοινή ευθύνη, για την πολλαπλή ευθύνη. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Αν θέλετε να βρείτε ποιος έχει την ευθύνη στην αλυσίδα αν υπάρχουν διάφορες επιχειρήσεις από διάφορες χώρες. Έτσι είναι στην Ευρώπη σήμερα. Σε οικοδομικές επιχειρήσεις, για παράδειγμα, έχετε ανθρώπους από πολλές και διαφορετικές χώρες, επιχειρήσεις από διαφορετικές χώρες. Ε, πρέπει να έχει κάποιος την ευθύνη στην αλυσίδα, να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνο γιατί. Ώστε όσοι δουλεύουν, να δουλεύουν κάτω από συνθήκες και αυτοί που παραγγέλνουν το χτίσιμο μιας οικοδομής, για παράδειγμα, έχουν την ευθύνη το ότι όντως οι εργάτες τους δουλεύουν κάτω από συνθήκες. Το έχουμε ξαναπεί και από πέρυσι, αλλά δεν είδαμε τίποτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει τον κανόνα της εσωτερικής αγοράς και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, στην Νορβηγία για παράδειγμα, υπάρχει αυτή η κοινωνική ευθύνη ή αυτή η αλυσιδωτή ευθύνη. Τροπολογία μας αριθμός 90 τώρα. Και 26. Και 86. Τι λέμε. Δεν λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σωστή προσέγγιση. Λέμε όμως ότι επί τόπου υπάρχει το πρόβλημα. Μπορεί η διατύπωση στις νομοθεσίες μας να είναι πάρα πολύ καλή, αλλά στην πραγματικότητα δεν γίνονται τα πράγματα όπως πρέπει. Και γι' αυτό θέλουμε να βελτιωθούν οι επιθεωρήσεις, η παρακολούθηση των δρόμενων επιτόπου, γιατί αλλιώ δεν έχει νόημα η καλή διατύπωση. Δεν κατηγορούμε δηλαδή ότι η νομοθεσία δεν είναι καλή, λέμε ότι αυτό που δεν γίνεται καλά είναι αυτό που γίνεται επιτόπου στο χώρο εργασίας. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε να συζητάμε τα προβλήματα που προκύπτουν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, ούτε πρέπει να φοβόμαστε να προχωράμε σε λύσεις. Για τελειώς η ξενοφοβία θα ενισχυθεί περισσότερο στην Ευρώπη. Και τότε οι άνθρωποι θα τσακώνονται μεταξύ τους, θα αγριεύουν όλο και περισσότερο, θα κρατάνε τους ξένους μακριά και δεν είναι αυτό που θέλω εγώ. Για να το αποφύγουμε λοιπόν Πρέπει να υπάρχει αυτή η αξιοπρεπή κινητικότητα και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, όχι μόνο στην νομοθεσία, αλλά και στην πράξη, στο χώρο εργασίας. Και αυτό είναι ο στόχος μας. Αυτό ζητάμε, αξιοπρεπή κινητικότητα. Μια τελευταία παρατήρηση τώρα. Ξέρω ότι μιλάω πολύ ώρα, αλλά έχω κάτι ακόμα που θέλω να σας διαβάσω πολύ σύντομα. Στο facebook μου πήρε ένα μήνυμα από έναν Ρουμάνο ο οποίο ενημερώθηκε για τις τη επιτροπή μας και ήθελε να μου διηγηθεί την ιστορία του. Είναι ένα νέος, 20 κάτι, και λέει 3 εκατομμύρια Ρουμάνοι δουλεύουν εκτός Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματα τα οποία δεν συζητιούνται ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε στα μέσα ενημέρωση. Ένα 22χρονο δούλευε, μάζευε κεράσια για 1000 ευρώ το μήνα δούλευε 6 μέρες τη εβδομάδα, 12 ώρες την ημέρα. Και τελικά, από ό,τι μου είπε, οι Ρουμάνοι τσακώνονται στις κερασιές, πραγματικά έρχονται στα χέρια με τους Πολωνούς. Και το ξέρω ότι υπάρχει αυτό. Και το ξέρω ότι συμβαίνει. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε, αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να ασχοληθούμε με τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν στους χώρους εργασίας και που έχουν να κάνουν με την κινητικότητα των εργαζομένων. Κατόπιν τούτων, πιστεύω ότι πρέπει να προωθήσουμε την κινητικότητα, να είναι πιο εύκολο για τους ανθρώπους να μετακινούνται και να δουλεύουν αλλού, αλλά να έχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα. Οι συντάξει, για παράδειγμα, και γενικότερα η προστασία. Παίρνω πάρα πολλά email σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Αυτά λοιπόν θέλω να προσταθούν στην έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κομφεράτη. Grazie Presidente. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τη... Ε, για όσα πρότεινε, ξεκινώντας από μια εκτίμηση την οποία συμμερίζομαι ότι η κινητικότητα στις χώρες της Ένωσης των εργαζομένων είναι κάτι το πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα θετικό να μπορούν να κινούνται ελεύθερα. Πρόκειται για μία από τις βάσεις της εσωτερικής αγοράς χωρίς να μπορεί κανείς να μετακινηθεί από τη μία χώρα στην άλλη χωρίς να βρει κατάλληλες συνθήκες εργασίες δύσκολα. Μήπως πιο σωστό θα ήταν να πω ότι μάλλον αποκλείεται η δυνατότητα πραγματοποίησης στόχων, αυτούς τους στόχους που έχει θέσει για το 2020 η Ευρώπη. Ε, μιλήσαμε και για ορισμένα δημογραφικά, από ηλικής πλευράς θα υπάρξουν δυσκολίες σε πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά ευνοούν μια φυσιολογική μετακίνηση που θα πρέπει βέβαια να ρυθμιστεί αλλά και να βοηθηθεί πρώτα απ' όλα. Ορισμένες τροπολογίες που υποβλήθηκαν είναι σημαντικές κατά την απόψή μου και τις οποίες σχολίασε ο εισηγητής να αναφερθώ σε πολύ λίγες ομάδες τροπολογιών ε, γύρω από τα θέματα της όλης συζήτησης. Πρέπει να καταρρύψουμε τα εμπόδια. Ένα από αυτά τα εμπόδια, λόγω των υλικών συνθήκων, για την ίση αμοιβή, ας πούμε, για ίση εργασία, αποτελεί μια από τις αφετηρίες της απαραίτητες. Το άλλο είναι τα δικαιώματα ανάμεσα σε αυτούς που εργάζονται και που δεν είναι τα ίδια δικαιώματα στις χώρες της Ένωσης. Όταν μιλάμε δε για δικαιώματα δεν θα πρέπει να σταματάμε στο στην σημαντική διάσταση των δικαιωμάτων ε, για την εργασία. Εντάξει, θα πρέπει να και για θέματα ηθαγένειας ε, θα πρέπει και εκεί να υπάρχει ισότητα. Μιλάμε για άτομα που εργάζονται σαν εργαζόμενος. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε αντικειμενικά τον εργαζόμενο από τον πολίτη και δεν μπορούν να δημιουργούνται συνθήκες ομοιόμορφες στην εργασία από τη στιγμή που να μην υπάρχει και για τους πολίτες μία ισότητα στην καθημερινή τους ζωή σαν πολίτες, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν κατά την απόψή μου είναι κάτι το πολύ σημαντικό η ανάλυση των ε, τροπολογιών και να λάβουμε υπόψη μας ταυτόχρονα αυτές τις διαπαιτήσεις για τον πολίτη και τον εργαζόμενο. Ανάμεσα στις ηλικές συνθήκες που και περισσότερο μας δημιουργούν δυσκολίες, δυσκολίες και στη γεννητικότητα είναι το εξή. Όχι μόνο η εργασία, τι γίνεται στο τέλος της δουλειάς. Ε, η πρόνοια είναι αποφαστική σημασία η φροντίδα. Θα πρέπει όσοι μετακινούνται όχι μόνο προς τα κοινά τίνουμε δηλαδή εντάξει τα ίδια μέτρα να ισχύσουν αλλά να μπορέσει κανείς να μεταφέρει μαζί του τη δική του μικρή κληρονομιά, τα δικαιώματά του, του μετά όσα έχει υποτιστεί και ίσως τελικά όμως δημιουργηθεί ένα φαινόμενο αρνητικό μάλλον. Υπάρχουν κάποιοι που εργάζονται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά θέλουν να επιστρέψουν σπίτι τους. Εντάξει, καλό, νόμιμο, σωστό. Εάν όμως δεν μπορούν μαζί τους ε, να φέρουν αυτά με τα οποία έχουν ποτιστεί όπως είπαμε και είναι τότε καταδικασμένοι να παραμείνουν στο τελευταίο τόπο εργαστήριο του πέρα από τη θέλησή του. Εκτό θέλησή του. Άρα λοιπόν αυτό για τη φροντίδα, για την πρόνοια, όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατάλληλα και είναι σημαντικά τόσο τουλάχιστον όσο και τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται, τα οποία γεννιούνται, τα οποία δημιουργούνται, όπω για κάποιον που εργάζεται εκεί σε αυτήν την εργασία. Κάτι το τελευταίο έχει να κάνει με τις κυρώσεις. Ε, πιστεύω ότι είναι και θετικό και αποτρεπτικό. Δηλαδή τα θετικά πρέπει να επιβραβεύονται και να υπάρχουν κυρώσει για τις αρνητικές ενέργειες. Εντάξει, το σύστημα προχωράει, μερικές φορές υπάρχουν και αποτελεσματικές ενέργειες, αλλά χρειάζεται, επαναλαμβάνω, όσοι δεν τηρούν τους κανόνες θα πρέπει να τιμωρούνται. Ακόμα περισσότερο σε ένα σύστημα το οποίο είναι σε αυτή τη φάση ανάπτυξης, αλλά για πολλά σημεία, για πολλές πτυχές ε, είναι και πειραματικό ακόμα. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Και δίνω το λόγο στην κυρία Κορνέλσεν. Τώρα έχετε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Υπάρχει το ερώτημα το οποίο έθεσε ο εισηγητής και το οποίο το αντιμετώπισε ήδη η κυρία Τούρουνεν. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εδώ είναι να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μοναχα μία ένωση οικονομιών, είναι μία ένωση ανθρώπων και η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων θα πρέπει να αποτελεί ένα δικαίωμα το οποίο να την χάνει παραβιάσεως μόνο αν είναι απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο. Και αν υπάρχει από χρόνο λόγος ο οποίος μπορεί να καταδειχθεί. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξει και ισότητα ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός προς τα κάτω μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων. Σε μία ενιαία αγορά υπάρχουν πολλές δυνατότητε για ένα κράτος μέλος να ανταγωνιστεί τους γειτονές του και τις άλλες χώρες σαν έδρα εγκατάστασης ε, μιας επιχείρησης, παραδείγματος χάρη. Επειδή όμως αυτά τα πλεονεκτήματα δεν είναι τόσο ισχυρά όσο ήταν στο παρελθόν οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν χρησιμοποιούν το κοινωνικό dumping τα κράτη-μέλη για τον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Θέλω να τονίσω επίση τη σημασία του να πούμε και κάτι σε σχέση με τα απαραίτητα μεταβατικά μέτρα. Δεν νομίζω ότι αυτά τα μεταβατικά μέτρα που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα ότι έχουν, δώσει, <clears throat> έχουν αποδώσει καρπούς και έχουν οδηγήσει σε πραγματικά ζωφερά αποτελέσματα σε ορισμένα κράτη-μέλη, υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων, ακόμα και μορφές δουλείας. Την 1η Μαΐου για όλες τις χώρες του 2004 τελικά θα αρθούν όλα αυτά τα μεταβατικά μέτρα, αλλά δεν θα ε, αρθούν για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και το δικό μου κρατός μέλος προς μεγάλη αμηχανία μου ανακοίνωσε αυτή τη βδομάδα ότι θα διατηρήσει τους φραγμούς για την εργασία Βουλγάρων και Ρουμάνων στην, στην ε, Ολλανδία και θα τους κάνει ακόμα πιο υψηλούς αυτούς τους φραγμούς. Αυτοί λοιπόν που έρχονται για να μαζέψουν μπανάνες από τη Ρουμανία στην Ολλανδία για πέντε χρόνια δεν μπορούν πια να το κάνουν και θα προτείνω και μια τροπολογία στην Ολομέλεια για να αντιμετωπιστεί αυτό το ειδικό θέμα. Κάτι ακόμα με την ε, ένταξη της Κροατίας που θα είναι στη νημερίσια διάταξη τον επόμενο χρόνο. Είμαι σίγουρη ότι κάτι κράτη-μέλη μεταξύ των οποίων και η Ολλανδία θα αποφασίσουν για εσωτερικούς λαϊκιστικούς λόγους να προτείνουν μεταβατικά μέτρα και για τους Κροάτες εργαζόμενους. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα και δεν έχει καμία χρησιμότητα γιατί η Κροατία έχει μόνο 3 εκατομμύρια κατοίκους, είναι σχετικά εύπορη χώρα σε σχέση με άλλες χώρες οι οποίες έγιναν πρόσφατα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι κάτι το παράδοξο περιλάβουμε λοιπόν και μια καταδίκη αυτής της ε, δυνατότητας και να κάνουμε ήδη μια έκκληση να μην γίνει πραγματικότητα κάτι τέτοιο. Επίσης είναι απαραίτητο να σταθούμε και στην αναγνώριση των γάμων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά υπόκειται στην επικουρικότητα. Δεν σημαίνει ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δεχθούν τους γάμους ατόμων του ίδιου φύλου. Ωραίο θα είναι αυτό, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα θέμα επικορικότητας. Απλώ σημαίνει ότι θα πρέπει να αναγνωρίζουν τους γάμους ατόμων από το ίδιο φύλλο. που έχουν συναυτεί σε κράτη-μέλη που έχουν γάμους ατόμων του ίδιου φύλου. Αν ένα σευγάρι Ολλανδέζων λεσβιών θέλει να χρησιμοποιήσει την ελεύθερη κυκλοφορία ε, των εργαζομένων, θα πρέπει η σύντροφό του να μπορεί να αναγνωρίζεται και σε άλλα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν γάμου ατόμων του ίδιου φύλου. Τέλο, ζητούμε από τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα τη διάκριση που υφίστανται άτομα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε άλλε χώρες μέλη. Στην ε, Ολλανδία, οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι και οι Πολωνοί όλοι αντιμετωπίζονται ω Πολωνοί. του. λένε Πολωνούς έτσι κι αλλιώ και είναι αντικείμενα σοβαρών διακρίσεων γιατί είναι αντικείμενα μιας στερεότυπης περιφροντικής μεταχείρισης. Και αυτό το θέμα δεν αντιμετωπίστηκε επαρκώς από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα καταθέσω την τροπολογία 68 για το θέμα αυτό και ελπίζω να με υποστηρίξετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κορνέλσεν. Και τώρα για να κλείσουμε τον γύρο αυτό, η κυρία Άκεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Χάρκιν. Και συγγνώμη ζητάω από τον εισηγητή που έλειψε από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του. Έπρεπε να πάω στην Επιτροπή Αναφορών, βλέπετε. Υπάρχουν και εκεί δικαιώματα των πολιτών. Ευχαριστώ πάντως τον εισηγητή έτσι καλώς για την έκθεσή του. Και έχω και μερικά σχόλια και ορισμένες ερωτήσεις. Συμφωνώ με τους πράσινους και με πολλά από τα σχόλιά τους όταν μιλάνε για την αξιοπρεπή κινητικότητα, όπως μιλάνε και για την αξιοπρεπή εργασία. Μακάρι να βρούμε τον τρόπο να τα περιγράψουμε αυτά. Όπως επίσης συμφωνώ και με την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ και της ξενοφοβίας. Σίγουρα με τροπολογίες θα πετύχουμε πολλά. Αλλά μπερδεύομαι λίγο για το θέμα αυτό της αναγνώρισης ε, ζευγαριών ε, του ιδίου φίλου που πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και σε άλλες χώρες που δεν αναγνωρίζουν τέτοιους γάμους. δεν ξέρω εδώ πέρα πώς μπορεί να γίνει. Αλλά από ό,τι θυμάμαι από την τροπολογία των Πρασίμων μιλάει για του ίδιου φίλου γάμους ή σχέσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο καινούργιε χώρε έχουν ή δεν έχουν προβλέπου κάτι τέτοιο. Πάντως, αυτό για να μου το εξηγήσετε. Και μερικά σχόλια. Και εγώ και ο κ. Γιώβενε, συναδελφός μου, έχουμε υποβάλει τροπολογίες για την αναγνώριση προσόντων, επαγγελματικών προσόντων και διπλωμάτων. Φαντάζομαι να τις δεχτεί ο εισηγητής. Για το θέμα των μεταβατικών μέτρων τώρα, που έχουν συζητηθεί εδώ, κάποιες τροπολογίες θέλουν να διαγράψουν κομμάτια που αναφέρονται σε εργαζόμενους από άλλες χώρες που συνεισφέρουν θετικά στην οικονομία κτλ. Εγώ δεν θα το ήθελα. Ανεξάρτητα από τα μεταβατικά μέτρα, αν οι χώρες μέλη έχουν λόγο να εφαρμόσουν τέτοια μεταβατικά μέτρα, δεν πρέπει να τα καταδικάζουμε. Μπορεί να μην συνάδει αυτό με το πνεύμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, αλλά παρόλα αυτά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε τις χώρες μέλη και όχι να τους επιβάλλουμε ε, να μην ε, έχουν μεταβατικά μέτρα. Γι' αυτό και δεν συμφωνώ με αυτό που λέει ότι οι χώρες που έχουν εφαρμόσει μεταβατικά μέτρα αυτό δεν είχε αρνητικές συνέπειες κτλ. Τροπολογία 26 των Πρασίνων. Τη διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή. Μιλάει για την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, ότι είναι θεμελιώδης ελευθερία. Ωραία. Και μετά λέει θέλει να υπάρχει σωστή προσέγγιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανάγκη μια προσέγγιση Ευρωπαϊκή Ένωση βασισμένη στα δικαιώματα για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Αν μιλάμε μόνο για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, μπορεί εδώ να διαπιστώσετε ότι το ίδιο μπορεί να ζητήσουμε και για την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και αγαθών. Και αν δούμε τι περιπτώσει έχουν πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η περίπτωση εκείνη που είχε να κάνει με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και το δικαίωμα στην απεργία. Υπάρχει κίνδυνος να μην υπάρχει συμμεταχείριση στα δικαστήρια. Εγώ φοβάμαι ότι υπάρχουν αρνητικές συνέπειες που δεν τις θέλουμε εδώ. Δεν είμαι εμπειρογνώμων. Θέτω το ζήτημα απλώς και νομίζω ότι πρέπει να το κοιτάξουμε προσεκτικά. Υπάρχει μια καλή τροπολογία που ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει ένα βαθμολόγιο για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε άλλη χώρα από τη δικιά τους. Να συγκρίνουμε δηλαδή τι συμβαίνει στα διάφορα κράτη-μέλη. Θα ήταν χρήσιμο αυτό. Να το ξέρουν οι πολίτες που σκοπεύουν να μετακινηθούν. Για τα κοινωνικά ζητήματα εξαιτία της διεύρυνσης ε, τώρα που λέει μια άλλη τροπολογία. Υποστηρίζω τις τροπολογίες όπως είναι 95 που ζητάει από την Επιτροπή να δημοσιεύσει τα θετικά που απορρέουν από την κινητικότητα των εργαζομένων και μιλάει επίσης και για την ενημέρωση των πολιτών για τα θετικά από τη μετακίνηση αυτή. Όπως λένε και οι πράσινοι, πολλές φορές ακούμε μόνο τα αρνητικά ή τέλος πάντων ε, τα δυνητικά αρνητικά, ξενοφοβία κλπ. Να πούμε και τα θετικά. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για τη δουλειά του. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Άρκιν. Θέλω να χαιρετήσω την παρουσία μιας ομάδας από δημοσιογράφων από την περιοχή της Εστρεμαδούρας στην Ισπανία, γείτονες δηλαδή από την Πορτογαλία, γείτονες της Πορτογαλίας και είναι ε, καλεσμένοι του Αλόνσο Σέρκας που είναι και αυτός από την περιοχή αυτή. Καλώς ήλθατε λοιπόν και Και θα ήθελα και η κυρία Εσαϊά να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θέλω να πω ότι συμμερίζομαι την άποψη της κυρίας Χάρκιν και συμμερίζομαι και την άποψή της για την τροπολογία αυτή για τους γάμους ιδίου φύλου. Υπάρχουν 14 χώρες που έχουν νόμους για συμβίωση ε, ζευγαριών του ιδίου φύλου πέντε που έχουν το δικαίωμα γάμου σε αυτήν την περίπτωση και άλλες τέσσερις χώρες που δεν έχουν καμία απολύτως νομοθεσία για ζευγάρια του ίδιου φύλου. Η τροπολογία αυτή λοιπόν θα πρέπει να εξασφαλίσει θέλει να εξασφαλίσει την ίση μεταχείριση, αλλά νομίζω ότι δημιουργεί μια ακόμα πιο άνηση μεταχείριση. Τα ζευγάρια αυτά που έρχονται από χώρες που υπάρχουν τέτοια νομοθεσία, δεν ξέρω πώς μπορούν να εξασφαλίσουν τα κοινωνικά ωφελήματα σε μια χώρα που δεν υπάρχει καθόλου νομοθεσία για τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι το θέμα αυτό πρέπει να παραμείνει στο πλαίσιο της επικουρικότητας και υποστηρίζω λοιπόν τη γραμμή και του ΕΛΚ στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Εντάξει. Κλείνουμε με αυτό τον γύρο παρεμβάσεων. Είδαμε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, πολυπίκυλες σε σχέση με ορισμένα σημεία και το τελευταίο αυτό θέμα για τους γάμους μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Και έχουμε και ένα άλλο σημαντικό θέμα, το οποίο είναι ακριβώς το θέμα αυτό της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, των δικαιωμάτων τους τον αγώνα κατά του κοινωνικού dumping και πιστεύω ότι θα παρουσιαστούν τροπολογίες. Για όλα αυτά τα θέματα δεν ξέρω αν ο κύριος Ουγγουριάνου θέλει να πει κάτι ακόμα, να κάνει κάποιο τελικό σχόλιο για όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν εδώ. Έχετε το λόγο λοιπόν αν το επιθυμείτε. Για την τελική σας καταληκτική παρέμβαση. Σας ευχαριστώ πολύ και πρόεδρε. Ε, εντυπωσιάζομαι από τα σχόλια των συναδέλφων και είμαι ευγνώμων για όλα αυτά τα οποία ανέφεραν. Μία δήλωση αρχής, αν θέλετε, μπορώ να κάνω, που έχει να κάνει με αυτά που ελέγχθηκαν. Είναι μια έκθεση για την κινητικότητα. Το πρόβλημα αυτής της έκθεσης είναι η κινητικότητα και η κινητικότητα των εργαζομένων <clears throat> είναι ένα πρόβλημα που καλύπτει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, γιατί υπάρχουν ακόμα φραγμοί και αυτό είναι σκανδαλώδες, πιστεύω. Η συνάδελφος από τους Πρασίνους που ανέφερε τα θέματα της φραουλοσυλλογής στην ε, Ολλανδία δεν είναι μοναχά ένα μεμονωμένο φαινόμενο αυτό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να το λύσουμε σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ο κίνδυνος ότι θα φέρουμε μέσα σε αυτή την έκθεση άλλα θέματα, παράπλευρα, οι διαδικασίες που δεν ανήκουν με αυτή την προβληματική. Πρέπει να επιλύσουμε πρώτα το πρόβλημα της κινητικότητας της εργασίας. Αλλιώς θα μετατρέψουμε αυτή την εργασία, κάτι το οποίο δεν πιστεύω ότι θα ήταν σωστό και εφικτό, σε μια έκθεση για ζητήματα ε, δόγματος κοινωνικής ευμάρειας ή να φάμε τη δουλειά του συναδέλφων μας που ασχολούνται με συντάξει και άλλα τέτοια θέματα. Δεν μπορώ εγώ τώρα να αντιμετωπίσω όλα αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι, αλλά θα το κάνω και σε μελλοντικέ ε, συζητήσει. Κύριε Μπικεβιτσούτε, σωστά, είπε από την αρχή ότι το πρόβλημα αυτής της έκθεσης είναι ακριβώς η ανάγκη να αρθούν όλοι οι φραγμοί για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αναφέρθηκε και στον αρνητικό αντίκτυπο ο οποίος μπορεί να προκύψει από την μετακίνηση των εργαζομένων στις χώρες προέλευσης αυτών των εργαζομένων. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν χωριστεί. Πολλές χώρες στην Ανατολική Ευρώπη είναι γεμάτες από τέτοια οικογενειακά δράματα που έχουν αυξηθεί, αυξάνονται κάθε χρόνο με ορατό τρόπο. για την κυρία Τσούρουνεν. Το πρόβλημα το οποίο αναφέρει το θέμα της μετακίνησης, της απόσπασης καλύτερα των εργαζομένων, μπορεί να φαίνεται ότι συνδέεται με την έκθεση ένα διαφορετικό και δεν είναι αντικείμενο αυτής της έκθεσης. Και θα έχουμε και μια ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους αποσπασμένους εργαζόμενους το Σεπτέμβριο. Και δεν μπορούμε τώρα να το αντιμετωπίσουμε μέσα σε αυτή την έκθεση και προτού παρουσιαστεί η ανακοίνωση της Κομισιόν. για τον κύριο Κοφεράτη. Συμφωνώ ότι οι συνδίκες εργασίας και διαβίωσης δεν μπορούν να παραγνωριστούν όταν κάποιος δουλεύει σε μια άλλη χώρα που την έχει επιλέξει θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αξιοπρεπούς εργασίας και διαβίωσης. Δεν ξέρω τώρα επίσης αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των συντάξεων, αυτό το πολύ θέμα σε αυτή την έκθεση. Μπορούμε να το αναφέρουμε, αλλά δεν νομίζω μπορούμε να το λύσουμε σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ την κυρία Κορνέλισεν. Αυτό είναι το πρώτο δίλημά μας σε αυτή τη συζήτηση. Αυτά τα οποία είπε επίση η κυρία Χάρκιν ρίχνουν φως σε αυτό το πρόβλημα για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αν προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση θα μπούμε σε ένα νομικό τέλμα και δεν είναι εύκολο να βγούμε από εκεί. Γιατί αυτές οι τροπολογίες που αναφέρθηκαν μπορεί να έχουν αντιφατικό χαρακτήρα σε νομικό επίπεδο. Και επίσης Χαίρομαι για αυτό που αναφέρατε για την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την πρόθεση της Ολλανδικής κυβέρνησης να παρεμποδίσει την έλευση Βουλγάρων και Ρουμάνων εργαζομένων στην χώρα εργασίας της Ολλανδίας. Επίσης, πράγματι, η Κροατία, από ό,τι μπορούμε να προβλέψουμε, θα είναι το επόμενο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι γελίο να έχουμε και πάλι τα ίδια προβλήματα με την ευκαιρία της προσχώρησης Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να κλείσω... Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι την κυρία Χάρκιν για τις παρατηρήσεις της και για την τελευταία της παρατήρηση τώρα. η ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει στοιχεία σε σχέση με την τωρινή στατιστική απεικόνηση την, της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι αγορές εργασίας της Δυτικής Ευρώπης με την έλευση εργαζομένων από την Ανατολική Ευρώπη. Τα στοιχεία υπάρχουν και έχουν δημοσιευτεί, αλλά πρέπει να αναδημοσιευθούν με νέο τρόπο, ώστε να είναι πιο εύκολο να τα αντιμετωπίσει κανεί, να είναι πιο εύληπτα αυτά τα στοιχεία. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Αντίθετα με το μύθο που είχε διαδοθεί είτε στην Αγγλία είτε σε άλλες χώρες, ότι δηλαδή θα υπάρξει μία <clears throat> είσοδος των ξένων εργαζομένων που θα είναι αρνητική για την τοπική οικονομία, δείχνει η εμπειρία αυτή, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο αν δεν κάνω λάθος, 1% του ΑΕΠ οφείλεται στην έλευση των ξένων εργαζομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό δεν είναι αμεληταίο. Και επίσης το παράδειγμα της Ιρλανδίας, κυρία Χάρκιν, είναι ακόμα πιο λαμπρό. Η Ιρλανδία αντιμετώπισε αυτή τη μεγάλη πρόκληση όταν δεν έθεσε κανένα φραγμό για τους ξένους εργαζομένους. Και το εγχείρημα αυτό ήταν μια μεγάλη πτυχία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λεκύη Πρόεδρος. Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της συζήτησης. Θέλω απλώς να σας υπενθυμίσω δύο θέματα. Πρώτον, ότι στην επόμενη συνεδρίαση της 24 η 25 Μαΐου θα έχουμε και την ε, άποψη του εισηγητή για τις τροπολογίες και τις τροπολογίες συμβιβασμού του και ενδιαμέσως σας πενθυμίζω ότι η έγκριση θα γίνει στις 15 και 16 Ιουνίου και θα πάει στην Ολομέλεια τον Ιούλιο, εάν θέλει ο Θεός. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα λοιπόν το οποίο προβλέπεται για την έκθεση αυτή. Και νομίζω ότι έχει εξαντληθεί η μερισία διάταξη και μπορούμε να κλείσουμε εδώ τη συνεδρίασή μας. Σας υπενθυμίζω ότι αύριο στις 9 επαναλαμβάνονται οι εργασίες μας και θα έχουμε τις ψηφοφορίες και θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους αυτούς που έλαβαν μέρος στις συνεδρίες και τους διερμηνείς μας επίσης ευχαριστώ.